Ladies and gentlemen, please take your seats. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. This is this is my last uh, possibility to to speak to you from the podium. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να σας μιλήσω από το πρόεδρο γι' αυτό αισθάνομαι συγκλονισμένος ως απερχόμενος πρόεδρος της, της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία που είχαμε. Αρχιερεσίες του Προεδρείου. Σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες μας, θα πρέπει να διαπιστώσουμε απαρτία με βάση τον κανόνα 195. Υπάρχει απαρτία. Ποιες είναι οι υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Ο Πάολο. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να προτείνω την υποψηφιότητα του κυρίου Καζίνη που ήταν και μέχρι τώρα πρόεδρος της Επιτροπής Σταγματικών Υποθέσεων και πολύ θα θέλαμε να συνεχίσει να προεδρεύει στην Επιτροπή. Νομίζω ότι άλλες συστάσεις είναι περίδες. Άλλες υποψηφιότητες υπάρχουν. If no, I think that we can proceed by a vote of... Ωραία, τότε διαβοής παρακαλώ να εγκρίνουμε την υποψηφιότητα του κυρίου, την εκλογή του κυρίου Καζίνη. Πρόεδρε Καζίνη, Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπό μου. Μάλλον <laughs> σίγουρο ήταν, είχαμε ήδη κλείσει συμφωνία σχετικά, αλλά δεν ξέρω, είπες ε, δεν είμαι ταπεινόφρον να πω ότι είναι πραγματική αυτή η εμπιστοσύνη. Πραγματική πάντως ή πραγματική δεν ξέρω, αλλά θα προσπαθήσω να ασκήσω τα καθήκοντά μου σαν πρόεδρος σε αυτή την υπόλοιπη θητεία με κάθε δυνατή προσπάθεια γιατί στην Επιτροπή, η Επιτροπή που έπαιξε και παλιότερα κύριο ρόλο σχετικά με τα θεσμικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα η Επιτροπή μας παίζει ακόμα σημαντικότερο ρόλο, κυρίως όσον αφορά το θέμα της συνθήκης ε, της συμφωνίας που είναι αντικείμενο συζήτηση, αλλά και μια νέα αρχιτεκτονική, μια νέα δόμηση και που καθοδηγείται με έξυπνο τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας τις βάσεις, τα θεμέλια και ακριβώς με τους λόγους που ξέρουμε ότι οθούν την Ευρώπη δεν θα μακρηγορήσω πάνω σε αυτό, αλλά πρέπει να εκλέξουμε τους τέσσερις αντιπροέδρους. Και εδώ οι ομάδες θα πρέπει να μας πούν ποιοι είναι οι υποψήφοι. Πριν να ξεκινήσουμε πάντως, πριν να προχωρήσουμε στην εκλογή των αντιπροέδρων, να χαιρετήσω το νέα μέλη της Επιτροπής ε, σχεδόν όπως πριν. Ε, ο νέο, το νέο μέλος είναι ο Αντωνιώτσι, τακτικό μέλος, ο Ρέχα επίσης τακτικό μέλος. Εντάξει, για να συντομεύσω, δεν θα προχωρήσω. Βέμπερ επίσης, ε, Γιώργος Γκαρσία κλπ. Τακτικά μέλη. Νομίζω ότι έχω συμπεριλάβει όλους. Θα ήθελα να τους χαιρετήσω, να τους ευχηθώ καλή δουλειά. Και προχωράμε τώρα στην εκλογή των αντιπρόεδρων. Μήπως υπάρχουν υποψηφιότητες λοιπόν σχετικά με τον πρώτο αντιπρόεδρο. Ε, εντάξει, εντάξει, κατάλαβα. Συγγνώμη από το συνάδελφο Γκουαλτιέρη που ήταν ήδη μέλος, αλλά... Όχι. Μέλος ή όχι μέλος πριν. Δεν ακούμε την απάντηση. Όχι, να μην τον αγγείλω. Δεν τον αγγείλω, λοιπόν. Ε, εντάξει, εντάξει. Ε, Τέλο πάντων, αυτό το λάθο δείχνει και τι σχέσει μα. Λοιπόν, ε, εκλογή αντιπροέδρων και για του σοσιαλιστέ. Ποιο είναι ο υποψήφιο, Η ομάδα μου θα προτείνει την κυρία Γκουρμάη ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Η υποψήφινο θα πρέπει να γίνουν δεκτή η κυρία Γκουρμάη απούσα σήμερα, αύριο παρούσα. Από την Ικαράγουα, από την Κοσταρίκα έρχεται. Και έστειλε mail πάντως που μας αναγγέλει ότι αποδέχεται την υποψηφιότητά της. Κάποιος άλλος υποψήφιος, όχι. Άρα λοιπόν, για βοήθεια. ποιοι είναι υπέρ της υποψηφιότητα της κυρίας Γκουρμάη. Ναι, εντάξει, γίνεται δεκτή. Ο δεύτερος αντιπρόεδρος μας τώρα, από το ΕΛΚ, κάποιος υποψήφιος. Εκ μέρους του ΕΛΚ, θα ήθελα να προτείνω την ε, ε, υποψηφία της κυρίας Κωνστάς Γκρίπ. Άρα ε, λοιπόν μια και δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, η κυρία Γκρίπ, εντάξει διαβοής, εκλέγεστε. Σας παρακαλούμε, ελάτε εδώ στο βήμα. Τρίτος αντιπρόεδρος, Νταφ να προτείνω την υποψηφιότητα του κ. Μέσσερ Σμιτ ως αντιπρόεδρο. Ο κ. Μέσσερ Σμιτ, λοιπόν. Μέσσερ Σμιτ. Μέσσερ Σμιτ. Απόν και εκείνος. Όχι, εκεί, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ στη μέση, μέση, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, αποδέχεστε την υποψηφιότητα, ναι. Αποδέχεστε, ναι. Εντάξει, άρα λοιπόν διαβοής και ο επιψήφιος γίνεται δεκτή η υποψηφιότητά του και εκλέγεται. Έχουμε τον τέταρτο τώρα αντιπρόεδρο. Ο Σεραφός Φατχόσκι. Στα ε, ονόματι της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των πολιτικών ομάδων θα ήθελα να προτείνω την υποψηφιότητα της κυρία... του κυρίου Φόξ. Κολέγα Φόξ. Ε. κύριος Φόξ λοιπόν. Απόν. Εντάξει όμως μας ειδοποίησε με mail, αποδέχεται την υποψηφιότητά του. Να δούμε λοιπόν. Για βοής. Ε, εντάξει εκλέγεται. Έτσι έχει λοιπόν η σύνθεση του προεδρίου. Και τώρα να περάσουμε στην ημερήσια μας διάταξη αυτή καθ' αυτή. Εγκρίνεται το σχέδιο ημερήσιας διάταξης που τις 17 Ιανουαρίου σας δόθηκε Σιωπή σας σημαίνει αποδοχή. Μενέντες Δεβίγκο, υφυπουργό για ευρωπαϊκές υποθέσεις στη χώρα του, και εισηγητή όμως ήταν για διάφορα θέματα σχετικά ας πούμε το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία με δύο σημεία που θα πρέπει να αποφασίσουμε είχε συντάξει μια πρώτη έκθεση, αλλά στη σημερινή μας ημερήσια διάταξη ήταν το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία, αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνει χωρίς να υπάρξει ένας αντικατεστάτης του εισηγητής. Αυτά λοιπόν και μετά θα δούμε. Θα τι αποφάσισαν, τι προτείνουν οι συντονιστές, αλλά το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να αφαιρεθεί και αναβάλλεται μέχρι να έχουμε τον νέο εισηγητή που θα εξετάσει το θέμα. Και αν συμφωνείτε θα έχουμε την έκθεση DAF για την προεκλογική διαδικασία και το πρωτόκολλο που η Δημοκρατία της Τσεχίας ε, ζητάει ώστε να προετοιμάσει τις αυριανέ πρωινέ ψηφοφορίες. Μέχρι τις 5.30 μάλλον από τις 4 μέχρι τις 5.30 4 μέχρι 5.30 με τη Δανική Προεδρία του Συμβουλίου Βάμεν Νίκολαη θα συνθούμε μαζί του και αύριο στο τέλος ακριβώς της ψηφοφορίας από τις 10.30 μέχρι τις 11.30 θα συναντηθούμε θα ακούσουμε την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Ευρωπαίο πολίτη και ο εκπρόσωπος ακριβώς της Επιτροπής θα μας ε, πει ποιος είναι το θέμα αυτό. Σοφή Μπέρναρτς που είναι αρμόδια τμήμα της Επιτροπής που είναι και υπεύθυνη για την Ευρωπαϊκή Χρονιά όπως ακριβώς έχει προγραμματιστεί το 2012, το γνωρίζετε όλοι σας. Και στις 11.30 αύριο το πρωί, μετά από τη σχετική ακρόση, θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών για το θέμα της ε, Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας δεν έχουμε τώρα άλλε παρατηρήσει από πλευρά τη Επιτροπή μα, εντάξει, το πρόγραμμα αυτό, το σχέδιο αυτό ε, με διάταξη εγκρίνεται. Να πάμε στι ανακοινώσει του Προέδρου. Τη 9 Ιανουαρίου στη συνάντησή μα οι συντονιστέ αποφάσισαν για τον συνάδελφο Ταρκόφσκι για την έκθεση για την αλλαγή των διατάξεων για τι γραπτέ δηλώσει σύμφωνα με το άρθρο 149 του κανονισμού. Προτείνεται λοιπόν αυτό να εγκριθεί στο σύνολό του και επίσης θεωρούν οι συντονιστές ότι για την Νομική Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς των υπαλλήλων θα πρέπει να δούμε το θέμα με το, θέμα αυτό. Και επίσης, συνάδελφος Ράγγελ, αντί για το Μενέντες Δεβίγκο, προτείνεται για την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου για την Ορλανδία, ακριβώ αντικαθιστώντας τον Μενέντες Ντεβίγκο που όπως σας είπαμε έγινε υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη χώρα του την Ισπανία. Αυτά. Αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, ισχύουν λοιπόν τα παραπάνω. Ναι. Ίσως κάτι που δεν άκουσα η Επιτροπή γιατί δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει για, το, για τους υπαλλήλους, γιατί θα πρέπει να έχουμε και μια γνωμοδότηση δική μας. Το θέμα είναι τόσο λεπτό και τόσο περίπλοκο που νομίζω ότι απαιτείται μια γνωμοδότηση δική μας. Δεν ξέρω, αλλά η αιτία άγνωστη σε μένα. Τι γίνεται, εδώ ο συνάδελφος Ταρκόφσκι πρόεδρευσε και γι' αυτό υπάρχουν τώρα μερικές δυσκολίες. Ο Νταφ, ο Νταφ όμως ο συνάδελφος Νταφ ήταν παρόν και ίσως θα μπορούσε να απαντήσει στο ερώτημά σου. Οι συντονιστές γιατί θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται μια γνωμοδότηση για την Νομική Επιτροπή για το καθεστώς των υπαλλήλων. Κύριε Νταφ. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη συζήτηση που έγινε, αλλά εκτιμήθηκε η ουσία της έκθεσης και καταλήξαμε στο ότι ε, ανέκυπταν συνταγματικά ζητήματα. Άρα καταλήξαμε στο ότι δεν θα έπρεπε να προετοιμαστεί σχετική γνωμοδότηση. Τέλο πάντων. Η Επιτροπή θα πάρει την τελική απόφαση. Απλά οι συντονιστές προτείνουν. Και ο Γκαργκάνη δεν ξέρω μήπως ε, ασέντησε κι άλλους που συμφωνούν με αυτόν να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων. Εγώ το είπα έτσι, αλλά αν μπορέσουμε να το συλλογιστούμε όλοι μαζί, καλό θα ήταν. Γκαλτιέρη. Ίσως να το σκεφτούμε κάπως για αυτό που λέει ο κύριος Γκαργκάνη και να μην αποφασίσουμε τώρα σε αυτήν τη συνάντησή μας, αλλά να αποφασίσουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Η Επιτροπή, εντάξει, οι συντονιστές υπέβλαν την πρόταση και αν θέλουν να επανέλθουν. Νομίζω εντάξει, απλό είναι. Για να το δούμε, να το δούμε στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών, λέει ο Πρόεδρος. Ένα ακόμα θέμα που θα συνακοινώσω είναι για τον προϋπολογισμό του 2012. Η Επιτροπή δική μας υιοθέτησε δύο τροπολογίες στην ε, πολιτική επικοινωνία με διάφορες δύο θέσεις στον προπολογισμό ουσιαστικά που θα έπρεπε να μπουν ε, στο αποθεματικό ε, μάλλον υπό επιφύλαξη κάτω γιατί διαπιστώσαμε διάφορες ελλείψεις, κάτι που δεν είχε συμπληρώσει η Επιτροπή ακριβώς. Και σαν προϋποθέσεις για να ε, ισχύσουν αυτές οι δύο θέσεις του προπλησμού είναι μια έκθεση πρότασης για τη διαχείριση των κοινών γραφείων ανακοινώσεων και το ανακοίνωση του προγράμματος εργασιών για το 2012. Επίσης, από πλευράς Επιτροπής, η παρουσίαση μιας στρατηγικής επικοινωνίας για τη διαθεσμική συνεργασία εν ώψη των ε, ευρωεκλογών του 2014. Ή τουλάχιστον οι ε, ερωτήσεις να γίνουν όσο γίνεται συντομότερα. Άρα λοιπόν προληπτικά σχετικά με την ε, πολιτική επικοινωνία σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και μετά την προετοιμασία ενός προγράμματος για τις ευρωεκλογές. Εντάξει, έχει τη διάθεση να το λύσει αυτό το πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γι' αυτό και ζήτησε μια συνάντηση με ορισμένα μέλη από την Επιτροπή μας που ειδικά ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό και για να διευκολυνθεί η επιτυχής διεξαγωγή αυτής της συνάντησης έστειλε τρία έγγραφα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα την έκθεση για την εφαρμογή των προτεραιοτήτων στην διαθεσμική ανακοινώσει για το 2000, από το 2010 και ακόμα ένα σχέδιο ακριβώς για το πρόγραμμα εργασίας του 2012 για τα κοινά γραφεία όπως είπαμε πριν και για την Ευρωπαϊκή Χρονιά Πολιτών μια πρόταση που θα εξεταστεί αύριο. Έτσι έχει κατάσταση, αυτή τη συνάντηση και οργανώνουμε, ειδικότερα το κάνει η γραμματεία και θα, ο κύριος Αντάργας θα ε, που είναι ο εισηγητή μα ε, για το 2012 και Γκουρμάη και Γκερέρο επίσης θα συμμετάσχουν οι συνάδελφοι που κατάθεσαν τροπολογίε ε, και οποιοδήποτε άλλος τώρα θα επιθυμούσε να συμμετάσχει να μας το πει. Μια συνάντηση για το θέμα των ανακοινώσεων της Επιτροπής και τις επαφές με διάφορα μέλη εδώ. Σημείο 6 έγκριση πρακτικών των συνεδριάσεων 21-22 Νοεμβρίου 2011. Τα έχουμε τα πρακτικά και όπως συνηθίζουμε ε, εγκρίνονται αυτά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αντιρρήσεις όπως και διαπιστώνουμε. Για τα 7 και 8 το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία σχετικά με την συνθήκη της Λισαβόνας σας είχα πει ότι σαν εισηγητής είχε οριστεί ο Μενέντες Δεβίγκο που όπως ε, είπαμε έγινε φυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θα πρέπει να τον αντικαταστήσουμε. Ο Σάνφος Ράγγελ προτείνεται από τους συναδέλφους ε, και αν συμφωνούμε όλοι μας τότε ο Ράγγελ είναι ο καινούριος συγγετής. Και όπως σας είχα πει και προηγουμένως ε, θα πρέπει πάντως να αφαιρεθεί από τη σημερινή από ημερήσια διάταξη. Και πάμε στο επόμενο σημείο για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που μας ε, απασχόλησε από το ξεκίνημα της θητείας μας και εμείς ε, και ειδικότερα τον συνάδελφο Νταφ ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε αύριο, γι' αυτό να τον ακούσουμε, να μας εξηγήσει ορισμένα πράγματα. Έχουμε, διαθέτουμε ακόμα λίγο χρόνο. Κύριε Νταφ, έχετε το λόγο. Yes, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επανερχόμαστε στο θέμα αυτό. Παρά το γεγονός ότι μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την προηγούμενη, μάλιστα, κοινοβουλευτική θητεία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει για υπερβολική σπουδή. Συζητήσαμε τη δεύτερη έκθεσή μου προηγουμένως και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε και πολύ επικοδομητική σύνθεση στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό τον Ιούλιο αλλά και η δεύτερη έκθεση ακολουθεί τη γραμμή της προηγούμενης μου έκθεσης που ήδη ήταν υπέρ μιας πανευρωπαϊκής εκλογικής περιφέρειας για την εκλογή 25 μελών από ε, πανευρωπαϊκούς ε, εκλογικούς, πανευρωπαϊκές εκλογικές λίστες και άρα ε, προτείνω μια ανακατανομή των εδρών για το 2014 λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τις δημογραφικές αλλαγές. Και σας μοίρασα και μία επιστολή. Ελπίζω να την έχετε λάβει όλοι. Με τα επίσημα δημογραφικά στοιχεία του 2000, για το 2012. Ο πίνακας λοιπόν που λάβατε είναι ενημερωμένος με τα νεότερα στοιχεία για το 2012. Και σε κάποια μέτρα φυσικά θα πρέπει να απαντήσουμε και στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν σε ό,τι αφορά την ε, αντιπροσωπευτικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ε, Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο εξέφρασε τέτοιες επικρίσεις. Και φυσικά είπαμε ανακατανομή των ε, δρών για το 2014 και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέοι Κροάτες βουλευτές μετά την προσχώρηση της Κροατίας τον Ιούλιο του 2013. Πάντως η ουσία της έκθεσης ε, ουσιαστικά κάνει μια επικαιροποίηση της κατάστασης. Και Αυτά γίνονται για να προετοιμαστεί το Κοινοβούλιο να, εκλέξει τον πρόεδρο τη Επιτροπή τον Ιούλιο πριν τι θερινέ διακοπέ. Προσπάθησα τη δεύτερη μου έκθεση να την κάνω πιο απλή, πιο συνοπτική και πιο συνενετική. Λιγότερο κατηγορηματική δηλαδή. Η έκθεση αυτή είναι πιο διαλλακτική ως προς τα σημεία που θα αποτελέσουν ε, ε, στοιχεία προς διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Για να δούμε τώρα εν συντομία τις συμβαστικές προτάσεις που σας έχω στείλει. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους συντονιστές και τους σκιώδεις ηγητές των ομάδων για την ε, ετοιμότητά τους ε, για συζήτηση και το διαλεκτικό τους πνεύμα. Η πρώτη συμβαστική πρόταση είναι η συμβαστική πρόταση Α και είμαι ευγνώμων όλος ιδιαίτερος προς τον κύριο Γουαλτιέρη ε, για την πρότασή του θέσπισης μιας νέας διαδικασίας στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την κατανομή των δρόμων. Ο κ. Γουαλτιέρη προτείνει και εγώ συμφωνώ μαζί του ότι η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών. Γιατί η απόφαση είναι πολύ σημαντική. Και θα πρέπει να προσπίζει τα συμφέροντα όλο, όσο περισσότερων μελών, κομμάτων και αντιπροσωπιών γίνεται. Η δεύτερη ε, συμβιβαστική πρόταση, η πρόταση Β, προσπαθεί να ικανοποιήσει εκείνους ε, που φρονούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή και να πάλι περισσότερα σε θέματα εσωτερικής ε, δημοκρατικής λειτουργίας των ε, κομμάτων και εντός των κρατών μελών. Ενώ άλλοι διαφωνούν. Ελπίζω να καταλήξουμε στη συμφωνία. Και η τροπολογία Γ είναι πολύ σημαντική γιατί εδώ ουσιαστικά θεσπίζεται ο διάλογος με το Συμβούλιο και αναφέρεται ρητά ότι στόχος είναι η, δράση, είναι η πράξη του 96 που για πρώτη φορά περιλαμβάνεται στο παράρτημα της έκθεσης και είπαμε ότι θέλουμε μια ε, γενική περιεκτική αναθεώρηση αυτής της πράξης που να καλύπτει πολλά σημεία. Πάντως αναγνωρίζουμε την ανάγκη επιτευξής συμφωνίας για όλα αυτά τα θέματα και όλος ιδιαίτερος για το θέμα του, της χρονικής στιγμής των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, ε, εφαρμογή το 2014 του συνόλου της πρότασης ή να υπάρξει καθυστέρηση για ορισμένα σημεία για αργότερα. Και αν, αν 25 ε, ευρωβουλευτές που θα εκλέγονται πανευρωπαϊκά θα πρέπει να περιορίζονται, να, να, ε, ε αφαιρούνται από τους 750 ή να προστίθενται στους 751. Και αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα επίμαχο. Και δεν υπάρχει συμφωνία προς το παρόν. Δεν έχει διαμορφωθεί μια κρατούσα γνώμη. Απλώς περιμένω να γίνουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για να αποσαφινιστεί κάπως το τοπίο. Και το τρίτο στοιχείο που καλούμαστε να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη είναι το σύστημα ψήφου για, τον για την πανευρωπαϊκή εκλογική λίστα. Αν θα είναι κλειστό το σύστημα ή, ε, ή μη κλειστό όπως προτάθηκε από μερικούς ε, συμπεριλαμβανομένου και μου. Η συμβαστική τροπολογία Δέλτα αναγνωρίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα αυτού του θέματος για όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τη διατύπωση αυτής της ε, συμβαστικής τροπολογίας <clears throat> ώστε να διαμορφωθεί μια αντιπροσωπευτική ε, ομάδα που θα διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις. Συμβαστική τροπολογία ε. Αναφέρει ε, ρητά τις αλλαγές της συνθήκης Λισαβόνας και στην ε, βουλευτική εντολή αλλά και για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον αντιπροσωπευτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια και εκπροσωπούνται άμεσα απευθείας οι πολίτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστώ τον Ρομπέρτο Γουαλτιέρη που υπέβαλε την τροπολογία γιατί ακόμη και οι ευρωβουλευτές δεν έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως τις αλλαγές που επιφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Η επόμενη συμβαστική τροπολογία συνδυάζει το ζωφερό στοιχείο της, του υψηλού ποσοστού της αποχής από τις ευρωεκλογές με το χρέος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το καθήκον του να προσελκύσει όλο και περισσότερους ψηφοφόρους στις κάλπες. Είναι σημαντικό να τονίσουμε αυτό το σημείο για να μην μας κατηγορήσει κανένας για συγκαταβατικότητα ως προς το πρόβλημα της μεγάλης αποχής από τις ευρωεκλογέ. Το σημείο G μιλά για την διακομματική δημοκρατία. Επίσης, το θέμα της ε, υπηκότητας και της ηθαγένειας αποτελούν το αντικείμενο της ε, επόμενης συμβαστικής τροπολογίας και εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ο ορισμός της εθνικότητας, υπηκότητας και της ηθαγένειας δεν είναι πάντοτε σαφή σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε άλλες χώρες ο ορισμός είναι σαφέστερος και σε άλλες λιγότερο σαφής. Και έχουμε και μία νέα διατύπωση για την ε, απαγόρευση ε, των διακρίσεων με βάση την ε, υπηκότητα για λόγους εθνικότητας. Τέλος, μετά από συνομιλίες που είχαμε τις ομάδες, αποφάσισα να αφήσουμε, να εγκαταλείψουμε την ιδέα της ε, μεταρρύθμισης, της αναθεώρησης και του πρωτοκόλου. Αλλά σε ό,τι αφορά την ακριβή διατύπωση των σκέψεων μας του πρωτοκόλου για τις ασυλίες ε, και τα προνόμια θα προκύψει μετά από διαπραγματεύσεις. Πάντως είχαμε πολλές διαφορετικές εμπειρίες σε ό,τι αφορά τη βουλευτική ασυλία μετά την συμφωνία που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το αρχικό παράρτημα 2 της έκθεσης μου. Είναι σημαντικό πάντως, ιδιαίτερα για τους πιο παλιούς ευρωβουλευτές, τους πιο παλέμαχους και τα πιο παλιά μέλη της Επιτροπής μας. θέλουμε να λάβουμε υπόψη και τις φρέσκες προτάσεις των νέων μελών. Πιστεύω ότι και κάποιες τέτοιες καινοτόμες ιδέες θα μπορούσαν να είναι επωφελείς για όλους. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι συμβαστικές προτάσεις που θα κληθούμε να ψηφίσουμε αύριο. Αυτά, ίσως μακρηγόρησα, πάντως σας ευχαριστώ για τη μέχρι τώρα τουλάχιστον υποστήριξη. Και τώρα συνάδελφος Σέφλιν έχει το λόγο. Αλλά παρακαλώ τον εισηγητή, τον κύριο Ντάφα, να συλλογιστεί πάνω σε ένα θέμα για τη συμβαστική τροπολογία Α με το άρθρο 231 για τον κανονισμό περί των λειτουργίας και ότι λαμβάνουμε την απόφασή μας με την πλειοψηφία των ψήφων των παρισταμένων, ενώ το άλλο είναι με την απόλυτη και είναι ουσιαστικά μια παραβίαση του άρθρου 231 της συνθήκες, μάλλον της συμφωνίας για την λειτουργία μας. Εντάξει, να το σκεφτούμε αυτό. διαπιστώνω όντως κάποια διαφορά από τη συνθήκη. Κάτι που σημαίνει ότι ως προς το σημείο αυτό θα πρέπει αντίστοιχα να τροποποιηθεί η συνθήκη. Πάντως υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία στην ε, έκθεση ε, μου που προϋποθέτουν ε, αναθεώρηση της συνθήκης σε ορισμένα σημεία. Πάντως κάποια στιγμή θα διαμορφωθεί ένα πλήρες πακέτο και αν συμφωνήσουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και αν υπάρξει και συμφωνία και εντό του Κοινοβουλίου, δεν νομίζω ότι το θέμα της αλλαγής των κανόνων ψηφοφορίας ε, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε, uh, thank you, Chairman, let me... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε για την επανεκλογή σας. Και να συγχαρώ φυσικά και τους αντιπροέδρους για την εκλογή τους. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ερμές μου ευχαριστής προς τον Άντριου Νταφ για την αγαστή συνεργασία που είχαμε για την έκθεσή του. φαίνεται σαν ένα από τα θέματα που θα απασχολούν συνεχώ την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων. Ε, ευελπιστώ όμω ότι θα δούμε και την μέρα τη διεκπαιρέωση αυτού του θέματο. Είχαμε εκτενέστατε διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό στο ΕΛΚ και τα μέλη του ΕΛΚ στην Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων είναι γενικώ υπέρ τη πανευρω... της πανευρωπαϊκής εκλογικής λίστας, αν και η πλειοψηφία του ΕΛΚ είναι μάλλον κατά έχει σοβαρούς ενδιασμούς. Και ως προς τη φόρμουλα που προτάθηκε, και εκεί υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες, γιατί φαίνεται ότι τα μεσαίου, μεσαίου μεγεθούς κράτη θα έχαναν ευρωβουλευτές. Βέβαια, με την προσχώρηση της Κροατίας κάποια ανακατονομή θα πρέπει να γίνει των εδρών. Εύλογο είναι, αλλά για τις 7 ή 8 μεσαίου μεγέθους χώρες είναι ε, αδιανόητο να χάσουν βουλευτικές έδρες τις οποίες θα πάρουν μεγαλύτερες χώρες. Είναι λογικό να μην ανεχθεί κάτι τέτοιο μια μεσαίου μεγέθους χώρα. Και είναι και αντιπαραγωγικό άλλωστε. Γιατί μια τέτοια φόρμουλα θα ενισχύσει τον ευρωσκεπτικισμό. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο. Τώρα για τις εκλογές ε, δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα. Τώρα για τις συμβαστικές τροπολογίες, για τη συμβαστική τροπολογία Δέλτα καταθέσαμε προφορική τροπολογία, για τη συμβαστική τροπολογία Ε. Είναι ενδιαφέρον το πώς διατυπώθηκε. Λέει, δεν εκπροσωπεί πια κατανάγκη μόνο τη χώρα από την οποία εξελέγει, αλλά ενδεχομένως εκπροσωπεί πολίτες από οποιαδήποτε χώρα κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ενδιαφέρουσες συνέπειες σε προεκλογική εκστρατεία και αλλού ή ε, στην πολιτική παρουσία. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί είναι γνωστό και στους 751 βουλευτές, αλλά δεν ξέρω πώς θα το αξιοποιήσουν και θα το εκμεταλλευτούν. Πάντως, όντως, νομικά εκπροσωπούμε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο τους συγκεκριμένους εκλογείς μας ή τη, τους συμπατριώτες μας. Τώρα, ένα σχόλιο για τη συμβαστική τροπολογία F. Σιγματάφη, για την ε, όλο και μεγαλύτερη αποχή από τις ευρωεκλογές. Θα πρέπει όντως να αντιμετωπίσουμε την ε, αδύρυτη πραγματικότητα της όλο και χαμηλότερης προσέλευσης των ψηφοφόρων στις κάλπες και θα πρέπει να βρούμε ε, μία λύση. Αλλά πρώτα να κάνουμε μία διάγνωση του προβλήματος. Ποια είναι τα αίτια αυτής της μεγάλης αποχής από τις ευρωεκλογέ. Ούτω ή άλλω, όλε οι εκλογέ δεν είναι μόνο σε ευρωεκλογέ που οι πολίτε ψηφίζουν λιγότερο. Και σε άλλου τομεί και σε άλλα σημαντικά θέματα ε, μειώνεται το ενδιαφέρον για την νομοθετική εξουσία η κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τα λόμπι. Φαίνεται ότι ε, δεν ε, ενδιαφέρονται. Θα πρέπει να δώσουμε την αξία του στην κοινωνία των πολιτών, στους εκπροσώπους, στα λόμπι, αλλά σε τελική ανάλυση η νομοθεσία και η ποιότητα της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι που θα φέρει πιο κοντά τους ψηφοφόρους στις κάλπες. Από εκεί θα, ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Πάντως ευχαριστώ Άντριου. Ήταν συναρπαστική όλη η διαδικασία για όλους μας και χαίρομαι που έλαβα και εγώ μέρος αυτή. Παρόλο που κράτησε πολύ. Ο κύριος Γουαλτιέρη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η θέση της ομάδας ακριβώς αυτής για την έκθεση DAF ή να το πω καλύτερα στην πρόταση για το ψηφοδέλτιο το πανευρωπαϊκό που αποτελεί και το κύριο σημείο είναι γνωστό αυτό σαν θέση. Γι' αυτό και δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με αυτό. Εμείς είμαστε υπέρ ενός ψηφοδελτίου πανευρωπαϊκού. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα λεπτό και ότι θα πρέπει να πετύχουμε μια ευρεία συνένεση στο κοινοβούλιο μας ε, για θέματα τα οποία αφορούν τις εκλογικές διαδικασίες ε, και την ίδια τη φύση αυτής ε, της λειτουργία της λεπτής που θα πρέπει, στην οποία θα πρέπει να συμμετάσχουμε και να προωθήσουμε. Χρειάζεται να επαναδιατυπώσουμε ή αναθεωρήσουμε, όπως το είπε και ο εισηγητής Νταφ, ώστε η έκθεση αυτή, η έκθεσή του, πέρα από μια έκθεση που αναφέρει διάφορες αρχές, να μπορέσουν όμως να αποτελέσουν ένα οδηγό, κάτι πιο ανοιχτό, καλύτερα από μια έκθεση που αφορά συγκεκριμένα πράγματα και προβλέπει και προτείνει. Είναι αυτή η διατύπωση, πιστεύουμε ότι ίσως είναι καλύτερη για να μπορέσει να πετύχει αυτή την πλατιά συνένεση που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό το, να το επαναλάβουμε, τόσο λεπτό θέμα και ευαίσθητο. Οι τροπολογίες, οι συμβαστικές, ε, θεωρούνται από εμά θετικές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Νταφ, ο οποίος και προχώρησε σε διάφορες ε, διορθώσεις σχετικά με την πρώτη διατύπωση αυτών. Θεωρήσαμε ότι αυτές οι διορθώσεις, τροποποιήσεις ήταν και οι κατάλληλες γιατί καθιστούν το κείμενο περισσότερο ε, μάλλον το καθιστούν καλύτερο ακριβώς ε, και μετά από διάφορες περικοπές από εδώ και εκεί και σχετικά με τη συμβαστική λύση Α και το θέμα που έθιξε και ο πρόεδρος για το πόσο είναι συμβατό αυτό με τις συνθήκες Ίσως στην περίπτωσή μας θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας προφορικής τροπολογίας και σύμφωνα με, γιατί δεν υπήρχε αυτό το θέμα αυτό το καθορίζει διαφορετικό από το προτείνει. Δεν ξέρω πώς καθορίζει κάτι που δεν μπορεί να καθοριστεί στα πλαίσια μιας ε, αναθεώρησης των συνθήκων. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε λοιπόν να αποτελέσει λύση στο πρόβλημα αυτό και σχετικά με το θέμα αυτό με το καθορίζει, προτείνει Ίσως ε, θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε και με την ημερομηνία των εκλογών. Εξακολουθώ να μην ε, με εξακολουθεί να μην με πείθει το ότι θα πρέπει ε, αυτή η έκθεση να προτείνει μία να, να προτείνει μια απόφαση για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Ίσως ένα κάποιο χρονοδιάγραμμα, αλλά όχι τίποτα περισσότερο. Άρα λοιπόν δεν με ικανοποιεί πάντα το ισχύον έξι άρθρο και νομίζω και προτείνω, δεν ξέρω, μήπως και οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ θα μπορούσαν να εξετάσουν ένα συνδυασμό ανάμεσα στην τροπολογία, αν δεν κάνω λάθος, 30 του συναδέλφου Βίλαντ και τη δικιά μου την τροπολογία που νομίζω ότι μπορούν να συνδυαστούν άνετα αυτή την 29. Για θα πρέπει να δω πάντα στον κατάλογο ψηφοφορίας. Για να δούμε τώρα και άλλα σημεία που με μπερδεύουν κάπως και θα πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικά σε σχέση και με τον κατάλογο ψηφοφορίας που προτείνει ο εισηγητής. Πάνω απ' όλα την τροπολογία 31 από πλευρά συναδέλφου Άγγλοντ. Ε, θυμάμαι μια μακρά συζήτηση που είχε διεξαχθεί εάν χρειάζεται να εισαχθούν έννοιες όπως αυτές της ε, εθνικής μειονότητας και μετά από μια λεπτή δύσκολη εργασία είχαμε πει τι ακριβώς ε, θεωρούμε, τι πιστεύουμε γι' αυτό για το μειονότητα πέρα από το εθνική που είναι κάτι το ιδιαίτερα λεπτό σαν θέμα λοιπόν ε, μπερδεμένο ε, είμαι γιατί βλέπω στην τροπολογία 31 αυτά που λέει εισηγητής και εύχομαι να έχουμε μία πλειοψηφία που θα απορρίψει την τροπολογία αυτή. Για την τροπολογία 35 για τους καταδικασθέντες εγώ το προτείνω και ελπίζω να τύχει θετικής αποδοχής και μετά και από πλευρά η τροπολογία, Χέφνερ η τροπολογία 20 επίσης θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Αυτό που βρίσκω εγώ σαν ερμηνεία στον άρθρο 2 είναι ότι αποτελεί ένα άρθρο που δεν μπαίνει στην ουσία αν χρειάζεται ή όχι μία αλλαγή του αριθμού αλλά έτσι σε μια πρώτη πρόχειρη ανάλυση νομίζω ότι είναι περιττή αυτή η τροπολογία. Δεν χρειάζεται τώρα αν αποτελεί προϋπόθεση για να πετύχουμε μια πλατύτερη συνένεση τότε η ομάδα μας εντάξει θα μπορούσε να το υποστηρίξει. Με ενδιαφέρει να ακούσω και την στάση των υπολείπων ομάδων σχετικά με το σημείο αυτό. Σε αυτά θα αρκεστώ το θέμα αυτό συζητήθηκε αρκετές φορές και γνωρίζουμε όλοι μας τα σχετικά επιχειρήματα. Και τώρα το λόγο έχει συνάδελφος Χέφνερ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ε, συγχαρώ για την επανεκλογή σας και εσάς και τους αντιπροέδρους. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή μας θα συνεχίσει να διέπεται από το πνεύμα συνεργασίας και αντικειμενικότητας, όπως και στο πρώτο τμήμα της θητείας άλλωστε. Βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση εξέταση της έκθεσης του Άντριου Νταφ. Νομίζω όμως ότι άξιζε τον κόπο. Δεν επαναλάβαμε δύο φορές τα ίδια πράγματα. Όχι, έγιναν πολλές συζητήσεις και μάλιστα επικοδομητικού χαρακτήρα και πολλά προέκυψαν από τις συζητήσεις αυτές. Η έκθεση αυτή μειώθηκε καθαρά ως προς τον όγκο της και νομίζω ότι αποτελεί μια καλύτερη βάση επί της οποίας μπορούν να συμφωνήσουν ακόμα και εκείνοι που είχαν αμφιβολίες στην αρχή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω και ότι πιστεύω ότι πλέον η έκθεση θα μπορέσει να βρει σύμφωνο μεγάλο τμήμα των συναδέλφων στο Κοινοβουλίο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την πολύ σημαντική και την πολύ καλή συνεργασία και θα πρέπει πάντα να συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τη δημοκρατία. Είναι ένα μεγάλο σφάλμα να θεωρούμε ότι έχουμε κατοχυρώσει τη δημοκρατία, το Κοινοβούλιο, το εκλογικό δίκαιο και ότι δεν χρειάζεται πλέον να τροποποιηθούν. Όχι, η δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο κατέχει κανείς, είναι κάτι το οποίο βιώνει κανείς και πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι απαραίτητο να τονωθεί και να αναπτυχθεί αυτός ο χαρακτήρας της δημοκρατίας. Με πιο σαφή τρόπο από ότι ως τώρα. Αυτό θα δώσει στους πολίτες την δυνατότητα να εκλέγουν υποψήφιους πέρα από τα το του εθνικού κράτους μέλους του. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα διεξάγεται με πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα οι ευρωεκλογέ και η σχετική προεκλογική συζήτηση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε και κοινέ πλατφόρμες για τους κοινούς αυτούς υποψηφίους. Νομίζω ότι πρόκειται για μια ευφύη προσέγγιση που δεν κάνει, αν θέλετε, ένα τεράστιο βήμα επί του παρόντος, αλλά προδιαθέτει για θετικές αλλαγές σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα του Ευρωκοινοβουλίου και των ευρωεκλογών. Αναφέρθηκε και προηγουμένω από τον συνάδελφο Αγχέλ ότι τα μεσαίας κλίμακας κράτη θα είναι αυτά που θα χάσουν. Αυτό το επιχείρημα προβλήθηκε πολλές φορές στην πρώτη συζήτηση. Πλέον δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουν με μεγάλη άνεση. Γιατί δεν ορίζεται ποιος ε, θα είναι, ποια θα είναι η σειρά για την ανάθεση των επιπλέον έτρων. Ορίζεται απλά ότι θα πρέπει να οριστεί ένα σχετικός τύπος. Τώρα θα πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία όχι για εκ νέου ορισμού όλων των στοιχείων. Ο κύριο Σόπλινγκ το είπε. Τότε κύριε Σόπλινγκ σας είχα καταδείξει ότι όταν πάρουμε μια γραμμική καμπή θα χάσουν τα μικρομεσαία, αν τα μεσαία κράτη. Αν δούμε όμως ε, μια παραβολική τέτοια γραμμή, δεν θα χάσουν οι μικρές, οι μεσαίες χώρες. Ο Άντριου Ντάφ το άφησε ανοιχτό αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον οποιοδήποτε σοβαρό επιχείρημα για να υποστηρίξει κανείς ότι τον βλάπτει το σύστημα αυτό. Θα πρέπει να βρούμε τη λύση αυτή από κοινού. Το ίδιο ισχύει, θεωρώ, και το θέμα του αντίκτυπου στην σημερινή κατανομή των εδρών. Και σε αυτό αναφέρεται η τροπολογία υπερθμών 20. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια προσφορά προς αυτούς που φοβούνται ότι οι διεθνικές έντρες πάντα και με προβλέψιμο τρόπο θα αποβαίνουν προς όφελος των μεγάλων κρατών και προς εις των μεσαίων κρατών και των μικρών κρατών. Νομίζω ότι με την τροπολογία αυτή καθίσταται σαφές ότι μπορεί να ακολουθηθεί μια διαδικασία για την ε, υποβολή υποψηφιών χωρίς να αλλάξει η φυστάμενη σύνθεση και κατανομή των εδρών. Να μην βλάπτεται και να μην ζημιώνεται κανείς αλλά να συμβάλλει έτσι στην, ε, στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό. Αυτό αποτελεί όρο από πλευράς μας. Και η προσφορά αυτή του Ρομπέρτο Γουαλτιέρη. Και θα δούμε κατά πόσο θα αποδεχτούν την προσφορά αυτή και οι υπόλοιπε ομάδε. Έχουμε εντωμεταξύ ανάμεσά μα τον Υπουργό για Θεσμικέ Υποθέσει ε, από πλευρά Δανική Προεδρία για το εξάμεινο αυτό. Ευχαριστούμε που ήλθε. Θα θέλαμε να οργανώσουμε τα πράγματα ως εξής. Διακόπτουμε τώρα τη συζήτηση για την έκθεση DAF για τον ενιαίο εκλογικό νόμο. Πολλά και διάφορα που θα πρέπει και να συζητήσουμε με την Δανική Προεδρία, γιατί όχι, και Τη συζήτηση αυτή θα την επαναλάβουμε γιατί έχουμε ακόμα μερικούς εγγεγραμμένους όπως την συνάδελφο Κούρμα και Στεραχάου και θα το κάνουμε σήμερα το απόγευμα αν έχουμε ακόμα χρόνο διαφορετικά την συνέχιση της συζήτησης θα την αναβάλουμε για αύριο το πρωί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον Υπουργό Νικολάη Βάμεν που ήδη στην αντιπροσωπεία στην Κοπενχάγη. Το Δεκέμβριο είχαμε συναντήσει, συναντηθήκαμε λοιπόν στην Κοπενχάγη, αν δεν κάνω λάθος, και συνάντηση των Προέδρων των Επίτροπων, ε, τι έχουμε συναντηθεί ήδη, και υπάρχει λοιπόν μια σχέση μεταξύ μας και τώρα τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε εμείς κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας είναι πολλά και διάφορα. Το θέμα που έχει να κάνει και είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή η συμφωνία που θα φτάσει στο Συμβούλιο Υπουργών προσεχώς, αλλά έχουμε και άλλα θέματα όπως την Ερευνητική Επιτροπή, το πρωτόκολλο σχετικά με τη δημοκρατία της Τσεχίας, με εισηγητή το συνάδελφο Νταφ, το νέο εκλογικό νόμο, το είπα αυτό, και για να είναι καρποφόρα αυτή η συνάντηση, εντάξει θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολλά και διάφορα, αλλά καλύτερα να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα των ερευνητικών επιτροπών με τον η Μάρτιν εισηγητή, απόντα σήμερα, άρα ο συνάδελφος Γκερέρο θα τον αντικαταστήσει, αλλά λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει στη συζήτησή μας είχαμε και μία, ένα διάστημα κάπως ε, συλλογισμού, ας το πούμε έτσι, για να δούμε καλύτερα τις θέσεις των κρατών μελών, των κυβερνήσεων, όπως και των κοινοβουλίων πάνω σε αυτό. Εντάξει, θα μπορούσαμε σήμερα από εσά να έχουμε τις απαραίτητες ε, λεπτομέρειες, τις πληροφορίες, μαζί με σας να αποφασίσουμε πώς θα οργανώσουμε τα θέματα αυτά. Από τη στιγμή που υπάρχει μια πραγματική διάθεση να φτάσουμε γρήγορα σε ένα αποτέλεσμα, γιατί θα μπει αυτό το θέμα, έχει οριστεί για την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου ή μήπως θα πρέπει να δούμε διαφορετικά τα πράγματα και να καθυστερήσουμε ακόμα ένα μήνα μέχρι να μπει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια, στην Μεσσία Διάταξη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για την εκλογή σας σε αυτή την ε, πολύ ωραία επιτροπή και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα θέματα που σας απασχολούν έχουν μεγάλη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσβλέπω σε πολύ στενή συνεργασία με την Επιτροπή σας. Επίσης, με, χαρά, ιδιαίτερη χαρά ξαναβλέπω τόσα γνώριμα πρόσωπα. Γιατί έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές και απόλαυσα ιδιαίτερα τη συνάντηση που είχαμε στην Κοπεχάγη. όπου είχαμε θίξει μερικά από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Μάλιστα, εκδηλώσατε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συζήτηση της έκθεσης Μάρτιν ε, της ε, Ερευνητικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εξεταστικής Επιτροπής. Τώρα να σας παρουσιάσω τη γενική προσέγγιση της ε, Δανικής Προεδρίας και μετά να ασχοληθώ με την έκθεση Μάρτιν. Όπως ξέρετε η Δανική Κυβέρνηση είναι σχετικά νεοσύστατη η νέα δανεική κυβέρνηση είναι πολύ φιλοευρωπαϊκή και το πρόγραμμά της το ίδιο και μάλιστα η ομιλία της Δανέζου Πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια α, το άδειξε αυτό. Και μάλιστα ε, η, είναι σημαντικό το γεγονό ότι έχουμε για πρώτη φορά σχετικά ε, αρμόδιο, υπουργό για τέτοια συνταγματικά θέματα δείχνει πόσο σημαντικό εκεί είναι για μας και η Επιτροπή σας. Και μάλιστα μία δραστήρια και ενεργητική προσέγγιση ως προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση φαίνεται και στην, στο γενικό πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εργασιών και να συμβάλλουμε και εμείς στην αντιμετώπιση μερικών τουλάχιστον από τις σοβαρότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως Προεδρία του Συμβουλίου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διεξαγάγουμε το έργο μας με επαγγελματικό και διαφανή τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι κλειδί για μια πραγματικά επιτυχημένη ε, Προεδρία μετά τη θέση ισχύ της συνθήκη τη Λισαβόνα. Εμεί φυσικά θα επικεντρωθούμε στην νομοθετική διαδικασία. Ο ε, Δανέζα Πρωθυπουργό ε, το επισήμανε αυτό στην Ολομέλη την προηγούμενη εβδομάδα και σας διαβεβαιώ ότι θέλουμε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα με απτές συνέπειες για τους πολίτες και να χειριστούμε αποτελεσματικά το πλήρες νομοθετικό πρόγραμμα που έχουμε ενώπιόν μας. Ε, το Κοινοβούλιο και οι ειδικέ επιτροπή συγκεκριμένα θα αποτελέσουν ζωτικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να αναζητήσουμε και να βρούμε συμβαστικές λύσεις στο Συμβούλιο, αλλά και μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά και ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε σε απτά αποτελέσματα. Αλλά ας είμαστε και ειλικρινεί. Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντα για όλα τα θέματα. Πάντως, ε, όπως προέκυψε και από με τις μέχρι τώρα συναντήσεις μας, πιστεύω ότι θα έχουμε μια σχέση εργασίας που ακόμη και όταν θα διαφωνούμε θα το κάνουμε με σεβασμό της γνώμης του άλλου και με πολύ επικοδομητικό τρόπο. Αυτή θα είναι η προσέγγιση της Προεδρίας και απέναντι στο Κοινοβούλιο και απέναντι στην Επιτροπή σας. Και φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε κι εσείς και αυτή θα είναι και αντίστοιχα η δική σας προσέγγιση απέναντι στην Προεδρία. Σε ό,τι αφορά τώρα την τη συμφωνία για τα δημοσιονομικά, μια και πρόκειται για δύο κυβερνητική συμφωνία, ε, το έργο, για το έργο αυτό δεν προεδρεύει η Ιδανική Προεδρία, γιατί η διαπραγματεύση γίνεται σε μια τυχό κομμάδα ε, και οι αποφάσει λαμβάνονται σε επίπεδο αρχικών κρατών και κυβερνήσεων. Και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει ηγετικό ρόλο στο θέμα αυτό. Όταν συναντηθήκαμε στην Κοπεχάγη στα τέλη Νοεμβρίου, είχαμε μια εκτενή συζήτηση ω προ την ανάγκη τη ε, αναθεώρηση τη συνθήκη για να εξασφαλίσουμε δημοσιονομική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, ε, ξέτασα ενδελεχώς και την ε, πρόταση του κ. Νταφ για πιθανή αναθεώρηση τη συνθήκη. Τότε βέβαια, τον Νοέμβριο, κανένα δεν μπορούσε να διανοηθεί την τραγωδία που θα ακολουθούσε το Δεκέμβριο, στις 9 Δεκεμβρίου, στη συνάντηση τη διάσκεψη κορυφή. Έγινε μια απόπειρα να βρεθεί λύση σε επίπεδο 27 χωρών, αλλά δυστυχώ δεν κατέστη δυνατό. Και δεδομένη στι οξύτε τη κρίση, η μεγαλύτερη πιτοραιότητα ήταν η εξασφάλιση τη ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα τη Ευρωζώνη. Ω εκ τούτου, 26 χώρε ε, αποφάσισαν να εφαρμόσουν ε, την απόφαση μέσω μια νέα διακυβερνητική συμφωνία. Σχεδόν όλε οι χώρε, ακόμη και η Δανία, προτίμησαν η απόφαση για την ε, δημοσιονομική σταθερότητα να περάσει από την διαδικασία αναθεώρησης συνθήκης, κάτι που προϋποθέτει συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω μιας διαδικασίας συντακτικής συνέλευσης. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Έχουμε παρόμοιες θεσμικές επιφυλάξεις για τη διακυβερνητική λύση. Και σας διαβεβαιώ ότι και εγώ μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 9 η Δεκεμβρίου έχω και εγώ σοβαρές επιφυλάξεις. Γιατί βλέπουμε ότι αν συνεχίσουμε τον κατακαιρματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγηθούμε σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, σε μια διάσπαση και σε μια πρόθεση της διακυβερνητικής μεθόδου αντί να πριτανεύσει η κοινοτική μέθοδος δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να βρούμε μια ιδεώδη λύση. Βέβαια κάναμε ό,τι, μπορέ, ό,τι μπορέσαμε και τουλάχιστον αποσοβήθηκε η χειρότερη κατάσταση. Και θέλουμε μια ρεαλιστική λύση για την ε, συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις διατράνωσαν με πολύ καλό τρόπο τα επιχειρήματά σας. Δεν θέλουμε να διασπαστεί η Ευρώπη σε δύο ομάδες αυτών το χωρών της Ευρωζώνης και το χωρών που είναι εκτός Ευρωζώνης. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν τέτοια χάσματα. Γι' αυτό και αναλύθηκαν προσπάθειες ώστε η συνεργασία για τη νέα συνθήκη να είναι συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία. Και στόχος μας είναι η νέα συμφωνία να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια στιγμή στο μέλλον. Τέλος, η νέα συμφωνία ανα, αναμειγνύει και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο σε πολλές δια, διατάξεις της συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εξασφαλίσει την συμμόρφωση με την συμφωνία αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσκαλείται στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και μάλιστα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από κάθε Συμβούλιο Κορυφής. Εγώ δεν, δεν ε, ε, συμφωνώ ότι η διακυβερνητική λύση είναι η ιδεώδης λύση, αλλά μετά την κρίση της 9ης Δεκεμβρίου ε, φάνηκε ότι όταν αντιμετωπίζουμε σοβαρότερες προκλήσεις μπορούμε με συνεργασία να βρούμε ρεαλιστικές λύσεις. Άρα φυσικά έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Εδώ έρχομαι μπροστά σας ως Προεδρία του Συμβουλίου και διαβεβαιώ ότι η Δανία θα υπογράψει την συμφωνία, τη συνθήκη και θα, συμφων... θα επιδιώξει συμφωνία και μεταξύ των χωρών εκτός Ευρωζώνης. Και θέλουμε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βρούμε λύση και στα εκκρεμή ζητήματα. Η νέα συμφωνία δεν θα επιλύσει όλα τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης, αλλά αποτελεί μια σημαντική συμφωνία πρόοδου και στόχο έχει να, να, να αποκαταστήσει μια διαρθρωτική ισορροπία, κάτι που θα συμβάλλει και στη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά θα συμβάλλει και στην εξηγήση των οικονομικών και στην προσπάθεια αποκατάστασης της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη, γιατί αυτές είναι οι πρωταρχικές προτεραιότητες της Δανικής Προεδρίας. Παρόλο που οι αποφάσεις της 9 Δεκεμβρίου δεν θα εφαρμοστούν μέσω μιας αναθεώρησης της Συνθήκης Εύρωσης, ε, Ένωσης, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν ε, μπροστά τους αναθεωρήσεις τη συνθήκη. Για παράδειγμα, έχουμε την αναθεώρηση συνθήκης σε σχέση με το Ιρλανδικό και το Τσεχικό πρωτόκολλο. Θα ήθελα να χαιρετήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να το επενέσω για την κατανόηση που έδειξε ως προς το αίτημα του Συμβουλίου να μην συγκληθεί συντακτική συνέλευση. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τη συνεργασία του ε, ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Βέβαια υπήρξαν κάποιες επιφυλάξεις προς το τσεχικό πρωτόκολλο. Πιστεύω πάντως ότι αν δεν ζητήσει κάτι διαφορετικό η τσεχική κυβέρνηση, θα πρέπει να τηρήσουμε την υπόσχεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Τσεχία ε, που δόθηκε το 2009 και, προβλέπει, και που επιτρέπει τη θέση σε ίσχυ της Συνδικής τη Λισαβόνα. Γνωρίζω ότι ένα από τα θέματα που ζητήσετε να εξεταστούν σήμερα είναι η έκθεση Μάρτιν στην Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και παρόλο που ο κύριος Μάρτη σήμερα δεν μπόρεσε να έρθει εδώ, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί έδειξε εμπιστοσύνη στην ε, Δανική Προεδρία για το χειρισμό αυτής της κατάστασης. Και για την ε, Ολομέλεια τον Εύριο, ε, ελπίζουμε να είναι ε, πραγματικά ενημερμένο ο διάλογο. και αυτή η προθυμότητα να συμμετάσχουμε στο διάλογο ε, εκτιμάται ιδιαίτερα και από το Συμβούλιο αλλά και από την Προεδρία. Να σα διαβεβαιώσω ότι η Ιδανική Προεδρία θα ανταποκριθεί με το ίδιο πνεύμα. Είμαστε από μια χώρα με έντονο κοινοβουλευτικό έλεγχο και με γνωστή παράδοση στη διαφάνεια. Μπορείτε λοιπόν να είσαστε απόλυτα βέβαιοι ότι στην Προεδρία του Συμβουλίου θα ξεκινήσουμε με ανοιχτό πνεύμα και με διάθεση να βρούμε λογικούς συμβιβασμού. Ωστόσο, όπως σας έχω δηλώσει και σε προηγούμενες, τελικρινή μεταξύ μας. Όπως σημείωσε το Νοέμβριο η Πολωνική Προεδρία, η έκθεση Μάρτιν ε, προκαλεί κάποιες σημαντικές αμφιβολίες από πλευράς του Συμβουλίου. Δυστυχώς, δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσουν ε, οι εργασίες σε τεχνικό επίπεδο μέχρι τις αρχές της Δανικής Προεδρίας. Άρα δεν θα είμαστε σε θέση να επισέλθουμε σήμερα σε λεπτομερή συζήτηση σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένε διατάξεις της έκθεση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ωστόσο για να απαντήσω σε κάποια προκαταρτικά θέματα τα οποία ενδεχομένως να τοπιστούν ως προβληματικά από το Συμβούλιο. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι σε τέτοια πρώιμη φάση δεν έχει δημορφωθεί ακόμα τοποθέτηση του Συμβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν ως ε, Προεδρία του Συμβουλίου, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε κάποιου τομεί όπου ενδεχομένω να υπάρχει διάσταση απόψεων για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία εξέβρεση λύσεων από κοινό. Θα χρειαστεί σκληρή δουλειά στο Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Αλλά αυτό είναι και το σλόγγαν μα για την Προεδρία. Europe at work, η Ευρώπη στη δουλειά. αυτό θα κάνουμε λοιπόν και σα διαβεβαιώ ότι θα δουλέψουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και βάλαμε την έκθεση Μάρτιν στις αρχές Ιανουαρίου ως μεγάλη προτεραιότητα και συζητηθήκαμε και με μέλη των κρατών μελών. Θα συζητηθούμε και με εκπροσώπους των κρατών μελών σήμερα, μετά από τη σημερινή ημέρη, μέρα. Και όπως ανέφερα ήδη στην Κοπενχάγη τον Νοέμβριο, σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμα πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και θέλουμε να συνεργαστούμε προκειμένου η Διευθυντική Επιτροπή να μπορέσει να αναλάβει το έργο το οποίο θέλει να αναλάβει. Θα ήθελα ωστόσο σήμερα να σας αναφέρω κάποιες προκαταρκτικές ανησυχίες οι οποίες εκφράστηκαν και που θεωρώ ότι θα είναι ε, σημαντικές και μπορεί να μας προκαλέσουν προβλήματα. Πρώτο θέμα. Υπήρξαν κάποιες ανησυχίες και από την νομική μας υπηρεσία σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής της έκθεσης σε ό,τι αφορά όλες τις αρμοδιότητες ε, που προτίθεται, που θέλουμε, που προτείνεται να δίνονται στην Διερευνητική Επιτροπή, σε ό,τι αφορά και το άρθρο 226 που αποτελεί τη νομική βάση. Ένα δεύτερο θέμα είναι το θέμα της συμμόρφωσης με τις αρχές της ανάθεσης Είναι σημαντικό το Συμβούλιο να διασφανίζει ότι οι αρμοδιότητες που θα χορηγηθούν και θα εκχωρηθούν στην Επιτροπή Διερευνητική δεν θα ξεπεράσουν αυτά που ορίζονται στις συνθήκες. Κατά τρίτον, εκφράστηκαν ανησυχίες για το πώς ε, στο σχέδιο προβλέπεται παρέμβαση και επέμβαση τη διερευνητική επιτροπή σε διάφορε διαδικασίε. Για παράδειγμα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης σε ποινική έρευνα. Και αυτό αρμόζει και συνάδει με το πλαίσιο του ε, άρθρου 226. Τουλάχιστον όσο συνεχίζεται η εξέταση μια ε, υπόθεση. Ε, Ξέρω ότι εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες για την πρόταση να εμφανίζονται σε μέλη της Επιτροπής ε, σε ακροάσεις χωρίς πρώτη έγκριση. Στο Συμβούλιο αυτό βρήκε σύμφωνες και τις αντιπροσωπείες. Κατά πέμπτον, ε, επίσης παρόμοιες αμφιβολίες για το κατά πόσο η Διερευνητική Επιτροπή θα έχει πρόσβαση σε τέτοια έγγραφα, ιδιαίτερα απόρριτα έγγραφα και κατά πόσο αυτό συνάδει με τη σχετική ε, νομοθεσία. Και τέλος εκφράστηκαν κάποιες αρχικές ανησυχίες σε ό,τι αφορά τις προτινόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ε, με τις ε, απαιτήσει τη Επιτροπή. Ε, σύμφωνα με την έκθεση Μάρτιν, θα πρέπει αυτά να κατοχυρώνονται στην εθνική νομοθεσία. Όλα αυτά είναι προκαταρτικά και δεν αποτελούν εξαντλητικέ αναφορέ και θα πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε στο μέλλον με πιο λεπτομερή τρόπο. Ξέρω ότι κάποιες από τις ανησυχίες βρίσκουν σύμφωνοι και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας την παρουσιάζω με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να διεξάγουμε έναν ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο προκειμένου να βρούμε, ελπίζω, λύσεις επί τις οποίες θα συμφωνήσουμε όλοι. Θεωρώ ότι δεν θα σας προκαλέσουν έκπληξη αυτά, καθότι είσαστε και εμπρεγνώμονες σε θέματα συνταγματικών υποθέσεων. Στην τελευταία περίπτωση τρία χρόνια πήραν οι διαπραγματεύσει προτού καταλήξουμε σε συμφωνία το 1995 και η έκθεση Μάρτιν θέτει κάποια από τα ερωτήματα που είχαν συζητηθεί εντελεχώ τότε. Νομίζω ότι σημαντικό είναι να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου τα θεσμικά όργανα να κάνουν μια ενημερωμένη συζήτηση για όλα αυτά τα περίπλοκα ζητήματα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε ως Προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει να συνενώσω και να καταφέρω να συγκεράσω τις απόψεις 27 κρατών μελών. Η εργασία αυτή μόλις έχει ξεκινήσει, ελπίζω, και εσείς συνάδελφοι και ω το Κοινοβούλιο να τα λάβετε αυτά υπόψη όταν θα αποφασίσετε για τα επόμενα βήματα εκ μέρου σας σε ό,τι αφορά και το χρονοδιάγραμμα. Να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία θα συνεχίσει να εργάζονται σκληρά για το θέμα αυτό τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, για να μπορέσουμε να προβούμε και σε πιο συγκεκριμένα σχόλια για την έκθεση και να αναφέρουμε τα σημεία που μας απασχολούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάρτιν για τη δουλειά του και για την προθυμότητά του να συνεργαστεί με το Συμβούλιο. Η καλή βάση συνεργασίας θα είναι χωρίς άλλο πολύ ωφέλιμη για την περαιτέρω συνεργασία μας. Θα ήθελα παράλληλα να πω ότι ως Δανός εκτιμώ ιδιαίτερα και σέβομαι την επιθυμία του Κοινοβουλίου να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα πρωτοβουλία στον τομέα αυτό για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία στο πλαίσιο των συνθήκων και θα ήθελα να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Και περνάω έτσι στην διατύπωση του κανονισμού 1049 για την πρόσβαση στα έγγραφα. Αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα για την Δανική, για την Δανική Προεδρία, γιατί η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική για την Ένωση και καθίσταται ακόμα πιο σημαντική με την ε, παραλευσή του χρόνου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εντός του Συμβουλίου και στο Κοινοβούλιο πολλές διαφορετικές απόψεις. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση. Οι διαπραγματεύσεις θα είναι σκληρές. Και καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν ευελιξία και προθυμία συνεργασίας. Ένα άλλο θέμα το οποίο ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στο άνοιγμα της λήψης αποφάσεων είναι η έναρξη της πρωτοβουλίας των ε, πολιτών τον Απρίλιο. Φυσικά η ΑΦΚΟ ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ στην όλη διαδικασία και οφείλουμε λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή και στην Επιτροπή σας. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ε, ευρωπαϊκής δημοκρατίας, γιατί επιτρέπει στο λαό της Ευρώπης, στους πολίτες της Ευρώπης να συμμετάσχουν ενεργά. Οι τεχνικές πτυχές ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες. Και ανυπομονώ να δω πώς η πρωτοβουλία των πολιτών θα γίνει αντιληπτή από τους πολίτες. Αποτελεί ένα εντελώς καινούριο κεφάλαιο στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Προσεγγίζουν έτσι οι πολίτες στην Ευρώπη. Όπως όλοι ξέρουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει η εποχή κρίση, αλλά θεωρώ ότι περνάμε και βασικά μια κρίση εμπιστοσύνη, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό έργο. Αυτό αποτελεί μια πρόκληση την οποία θα πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά και πιστεύω ειλικρινά ότι η πρωτοβουλία των πολιτών θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση και για να καταπολεμηθεί το έλλειμμα τη εμπιστοσύνη Αύριο έχω την τιμή να ξεκινήσω με τον ε, Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς στην Επιτροπή μια σχετική διάσκεψη. Ξέρω ότι πολλοί από εσά θα συμμετάσχετε και πραγματικά προσβλέπω σε αυτή τη συνεδρίαση. Αποτελεί η πρωτοβουλία των πολιτών ένα εξαιρετικό παράδειγμα των όσων ελπίζουμε να πετύχουμε στην Προεδρία μας. Ξέρω ότι πολλά θέματα θα πρέπει να συζητηθούν και δεν πρόκειται να συνεχίσω τα εισαγωγικά μου σχόλια. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η Ιδανική Προεδρία ε, απόλαυσε πραγματικά τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή σας και θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία με εσάς. Και στο πνεύμα αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε. Ελπίζω να είμαστε αποδοτική, αποτελεσματική στα αποτελέσματα που θα πετύχουμε για τους Ευρωπαίου πολίτες. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Ευχαριστούμε τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Πάνω σε αυτό το ειδικό σημείο, με διάφορα θέματα, το θέμα ακριβώς των ερευνητικών επιτροπών εκεί δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε, θα πρέπει να εξετάσουμε καλύτερα τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς δεν μας ζητείτε να κλείσουμε το θέμα μέχρι το Φεβρουάριο. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Ναι. Σχετικά με τα διάφορα θέματα που θίξατε εσείς, ξεκινάει η συζήτηση να ακούσουμε τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Συνάδελφος Ταρκόφσκι, θα πρέπει να αφήσουμε χρόνο όμως το τέλος τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για να απαντήσει. Γι' αυτό παρακαλώ το πολύ πέντε λεπτά ο καθένας. Ταρκόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και για την επίσκεψή σας και για το ανοιχτό πνεύμα σας. Εδώ είμαι εδώ. Για την ανοιχτή και διαλλακτική της προσέγγιση σε ό,τι αφορά το φορολογικό, το δημοσιονομικό συγγνώμη πακέτο. Φαίνεται ότι η Ιδανική Προεδρία ε, έχει για το δημοσιονομικό πακέτο παρόμοια προσέγγιση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον για τα πιο σημαντικά θέματα, δηλαδή την διασφάλιση, διαφύλαξη της κοινοτικής μεθόδου και την χρήση όσο γίνεται περισσότερο με ανάμειξη των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, αποφεύγοντας τις παράλληλες δομές και δεύτερο, η αποφυγή του κινδύνου κατακαιρματισμού ώστε όλο και περισσότερες χώρες να, να συμμετέχουν στην ε, λήψη των αποφάσεων. Γιατί ούτω ή άλλω το δημοσιονομικό πακέτο όλου μα θα μα επηρεάσει, άσχετα από το να κάνει ανήκει όχι στην Ευρωζώνη. Νομίζω ήταν θετικέ οι διαπραγματεύσει και είπατε ότι διαφαίνεται μια ρεαλιστική και απτή λύση. Μήπως προτρέχετε όμως κύριε Υπουργέ αναγγέλλοντας μια τέτοια πιθανότητα. Γιατί αυτό που έχουμε επιτάπητος, ιδιαίτερα μετά από ένα ενδιαφέρον και απρόβλεπτο ε, τρίτο σχέδιο που ε, έπεσε λίγο ως, ουρανός, ε, ως κεραυνός ενεθρία δεν βλέπω και πολλές θετικές εξελίξεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε αίσια έκβαση. Βέβαια είπατε ότι η Δανία πολύ ευχαριστώ υπογράψει τη συμφωνία και θα την εφαρμόσει. Μετά την διαθέτηση όμως των εκκρεμωτήτων είπατε τι ακριβώς εννοείτε, ποιες είναι οι εκκρεμότητες κατά τη γνώμη σας και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις θα ήταν πρόθυμη η Δανία να υπογράψει τη νέα συμφωνία. Είπατε επίσης ότι υπάρχει ο κίνδυνος, ότι ο κίνδυνος μάλλον για Ευρώπη δύο ταχυτήτων έχει αποσοβηθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το σύμφωνο είναι ανοιχτό προς συμμετοχή όλων και προσιτό σε όλους. Βέβαια αυτό δεν φαίνεται από το σημερινό κείμενο. Είπατε όμως ότι αναμένεται νέα εκδοχή και δεν είμαστε βέβαιοι για το περιεχόμενό της. Πάντως, ε, για τα πιο σημαντικά θέματα. Άρθρο 2. Εμείς ε, θέλαμε όσο, και μεγαλύτερη, όσο γίνεται μεγαλύτερη εφαρμογή της κοινοτικής μεθόδου και της ενισχυμένης συνεργασίας για τα νομοθετικά ζητήματα. θέλουμε αυτό το άρθρο να έχει κατηγορηματική διατύπωση. Βέβαια, δυστυχώς έχει αλλοιωθεί και ε, μιλάει για τις συνήθεις ε, διαδικασίες της συνθήκης. Εμείς θέλαμε μια πολύ πιο κατηγορηματική διατύπωση για να ε, τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν το μέτρο του δυνατού και περισσότερο την κοινωτική μέθοδο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμμετοχή των μελών της Ευρωζώνης. Τώρα, αυτό που έχουμε τάπητος με όλες τις επιφυλάξεις, μόνο άπαξ το χρόνο και μόνο όπου δει, δεν θα έλεγα ότι παρά είναι αισιόδοξε οι προοπτικές. Και για το σημείο αυτό και πάλι, ένα σχόλιο συναφές με την αναγγελία της υπογραφής της συμφωνίας από τη Δανία. Και τι γίνεται Κατά τη γνώμη σας, ε, ε, τι όροι θα πρέπει να συντρέχουν ε, ώστε να προσυπογράψετε και εσείς και να εφαρμόσετε το φορολογικό, το φορολογικό δημοσιονομικό πακέτο. Αυτά σας ευχαριστούμε που εστερνίζετε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για τις ερωτήσεις που σας έθεσα. Ναι, Γκερέρο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Έχουμε ήδη συναντηθεί κάποιες προηγούμενες φορές για να κάνουμε και ένα απολογισμό των διαφόρων υποθέσεων που θα εξετάσουμε εδώ στην Επιτροπή μας και είχαμε και μια συνάντηση ιδιαίτερα χρήσιμη και όσον αφορά το διάλογο και την όλη συζήτηση για τις διάφορες υποθέσεις επί της ουσίας. Χαίρομαι που η θέση της Δανικής Προεδρίας είναι να πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα στην φάση αυτή και θα ήθελα να μιλήσω για τρεις συγκεκριμένες διαφορετικές υποθέσεις ε, για τις ερευνητικές επιτροπές. Ε, ο Ντέβιντ Μάρτιν είναι Συγητή ε, και σε άλλες δύο και εντάξει πέρα από τη διακυβερνητική συμφωνία για τον Ρομπέρτο Κορατιέρη που θα εξετάσει αυτά, που θα αναφερθεί σε αυτά, γιατί θα ήταν προδοσία από μένα. Εκείνο είναι από τα μέλη του Κοινοβουλίου που διαπραγματεύτηκε στην ομάδα εργασία. Εντάξει, να προσπαθήσω εγώ να αντικαταστήσω σε ένα θέμα που γνωρίζει τα πράγματα πολύ καλύτερα από εμένα. Εδώ πρώτα απ' όλα να μιλήσω τι θα γίνει αύριο το πρωί ή και σήμερα το απόγευμα θα το δούμε. Αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε για τα πρωτόκολλα της Δημοκρατίας της Αιχίας και, της, και την Ιρλανδία. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σχετικά με την Ιρλανδία εδώ στην Επιτροπή μας. Θα πρέπει να δούμε όμως ε, για τα προβλήματα για το πρωτόκολλο της Δημοκρατίας της Αιχίας. Δεν ξέρω τώρα αν περισσότεροι υιοθετούν ή όχι μια ερμηνεία για το πρωτόκολλο που προωθείται από το Συμβούλιο για να υπογράψει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό είναι νόμιμο, δεν ξέρω και υπάρχει μια πρόταση του εισηγητού. Το Κοινοβούλιο το απορρίπτει και το Συμβούλιο όμως ε, το υιοθετεί. Θα πρέπει βέβαια να το τονίσουμε όπως το γνωρίζει καλύτερα από μένα η, προ... η Προεδρία στη Δημοκρατία της Αιχίας, εδώ στο Κοινοβούλιο υπάρχουν διαφορετικές αντιμετωπίσεις αυτού του θέματος. Να, δεν ξέρω εάν το Συμβούλιο επειδή είχε αναλάβει κάποτε κάτι απέναντι στο Πρόεδρο της Τσεχίας το Κοινοβούλιο θα ήθελε να δηλώσει ότι η συμφωνία αυτή όμως δεν σέβεται όπως πρέπει την δημοκρατική διαδικασία. Δεύτερη υπόθεση στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ δεν μίλησε για αυτήν ο υπουργό στα όσα είπε προηγουμένως είναι η, η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Συμφωνία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και είναι κάτι που έχει ολοκληρωθεί στα πλαίσια διαπραγμάτευσης από την Επιτροπή. Ορισμένες ε, αντίθετες απόψεις όμως υπήρχαν από το Συμβούλιο στα διάφορα κράτη-μέλη και ίσως θα έπρεπε να παροτρύνουμε, να προωθήσουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε μια συμφωνία, γιατί δεν θα μπορούσε κανείς να καταλάβει ότι θα αφήναμε μια ολόκληρη τη θητεία έτσι του Κοινοβουλίου να περάσει, χωρίς να ολοκληρωθεί αυτό και την εντολή για την ε, συνθήκη της Λισαβόνα, ώστε να προσυπογράψουμε εμείς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Συμφωνία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ακόμα για το θέμα των ερευνητικών επιτροπών. Δεν θα προσθέσω τίποτα ιδιαίτερο στα όσα είπε ο Υπουργός, αλλά τη μετάδοση του βασικού μηνύματος, τι γίνεται με την όλη συγκυρία. Και το βασικό μήνυμα ποιο είναι. Ο Κοινοβούλιο όπως αναγνώρισε και τόνισε την αξία του ο υπουργό είναι να προωθήσει αυτό το θέμα για τι ερευνητικέ επιτροπέ. Ε, αυτά τα μέσα που διαθέτει η Ερευνητική Επιτροπή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι κάπω ισχνές ε, για να μπορέσει να προχωρήσει στην έρευνα εάν είχαμε ή όχι μία, ένα σεβασμό στα όσα ε, υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και τώρα στο τέλος ε, για να δει κανεί τι ακριβώς έχει γίνει απλά και μόνο προχωράει σε συστάσεις αλλά δεν λαμβάνει αποφάσεις όμως ε, γιατί αυτές, αυτό είναι αρμοδιότητες άλλων οργάνων. Θα πρέπει να δούμε ίσως τις ίδιες αρμοδιότητες όπως και τα εθνικά κοινοβούλια όταν ακριβώς προχωρούν στη σύσταση ερευνητικών επιτροπών και εκείνες που ζητούν εκείνο που ζητούνται, ζητείται να παρουσιαστούν μπροστά σε αυτές τις επιτροπές, να μην μπορούν να το αποφύγουν. Όπως μου είπε ο κύριος Μάρτιν, παραμένει ε, ανοιχτός, εντάξει, και να καθυστερήσει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια, να αλλάξει η ημερομηνία από τη στιγμή που θα, όπως είπατε και εσείς, θα εκφραστεί μια διάθεση για ένα συνδυασμό απόψεων, να βρούμε λύσεις. Ε, εντάξει, πάντως να μην καθυστερήσει αυτή η ψηφοφορία πέρα από τον Απρίλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. τον Υπουργό βάρμεν να καλωσορίσω θερμά με και θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Έτσι και οι ευρωπαϊκές υποθέσεις ε, είναι μια θέση ιδιαίτερα σημαντική, κάτι το ιδιαίτερα θετικό. Να δούμε τώρα στο Fiscal Compact τι γίνεται. Χαίρομαι γιατί η δανική κυβέρνηση συμμερίζεται πολλές από τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, συνθήκη αυτή. Η θέση μας, όπως είναι γνωστό, είναι ότι απαιτείται αυτή η συνθήκη από θεσμικής πλευράς και νομικής πλευράς και αν ε, ρίξουμε μια ματιά στα διάφορα άρθρα δεν ε, βλέπουμε κάτι που θα απαιτούσε μία αναθεώρηση των συνθήκων. Τώρα ακριβώς που το άρθρο το 3 λέει ότι ο χρυσός κανόνας θα πρέπει να είναι ακριβώς περισσότερο το Σύνταγμα, κάτι που υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα από τη δική σας την κυβέρνηση. Και σίγουρα δεν θα διαφοροποιούσε ιδιαίτερα τα πράγματα στα πλαίσια μιας δευτερεύουσας νομοθεσίας. Το reverse qualified majority απορρίφθηκε αυτό από πολλές κυβερνήσεις που τα θέλουν ε, στην άλλη δέσμη και ίσως εκεί ακριβώς θα μπορούσε και το 8-2 για τις κυρώσεις για το δικαστήριο αυτό είναι συζητήσιμο ακριβώς ε, ε, τη συνάντηση της Δευτέρα το βράδυ φάνηκαν διάφορε ανησυχίε ε, τι γίνεται από νομική πλευρά για το άρθρο 8.2 και σας προσκαλώ να το συλλογιστείτε. Εάν χρειάζεται κάτι παρόμοιο, να αφήσουμε μια νομική παρόμοια βεβαιότητα, παρόμοιου Εύρου σε μια συνθήκη που δυστυχώς ε, έχει, πάρει, έχει παίξει ένα ρόλο και στην εκτίμηση των αγορών. Γι' αυτό σας παρακαλώ να επιμείνουμε πάνω σε αυτό. Πώς δεν θα πρέπει να συνδυάσουμε την ήδη ισχνή νομική βάση του 273 σχετικά με το πρώτο εδάφιο το 8, ακριβώς τον διατικό ρόλο του δικαστηρίου και μετά να ζητήσουμε το δικαστήριο να συνδυάσει κυρώσεις του άρθρου 260 αυτό δεν γίνεται κατά την απόψή μου σχετικά με μια διακυβερνητική συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντως, ε, παρόλες τις αμφιβολίες αυτές, ε, θεώρησε ότι θα πρέπει ιδιαίτερα να ασχοληθεί και μάλιστα επικοδομητικά με αυτό για να μειώσει τις ζημιές, ε, να τις να βελτιώσει κάπως ε, αυτά τα πράγματα στη συνθήκη και στη τελευταία συνάντηση ακριβώς ε, είχαμε διάφορα μικροβηματάκια προς τα εμπρός και το άρθρο 3 είναι σημαντικό που επισήμως έγινε δεκτό με την τροπολογία μας για αναφορά στην ε, ορολογία του six pack και αυτό το deficit επίσης είναι ε, μπήκε στο 0,5 αντί για 1, ακριβώς μέσω με διακυβερνητική, με διακυβερνητική οδό, αντί για την τακτική νομική διαδικασία. Εντάξει, εκ των υστέρων θα τα διορθώσουμε αυτό, γιατί αυτό είναι δεικτικό ότι κανένα κράτος μελός δεν ζήτησε το 0,5 στη συζήτηση για το 6-pack, Εκτός από μια εβδομάδα μετά που ίσχυσε ζήτησαν το 05 μέσω μια διακυβερνητικής ε, διάσκεψης παρακάμπτοντας την τακτική διαδικασία. Είναι κάτι το χαρακτηριστικό και μια σελίδα όχι και τόσο φωτεινή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κάτι ακόμα με μια συνένεση είναι η συμμετοχή στο Summit του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διευκρινίσω τα πράγματα που στα είπε ο Υπουργός, το maybe invited to be heard, το να προσκληθεί κανείς να ακούσει τα πράγματα και πώς έχει κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν ισχύει αυτό για μια άτυπη συνάντηση όπως είναι η συνάντηση του Eurosummit όπως το λέει το άρθρο 12 της συνθήκης και να έχουμε περισμούς διαδικαστικούς που θυμίζουν εκείνους τους περιορισμούς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι όμως θεσμικό όργανο. Έτσι, ε, δεν θα μπορούσε Κανεί νομίζω να χαράξει παρόμοια όρια από τη στιγμή πρόκειται για άτυπε συναντήσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα λήψεω αποφάσεων. Αναφέρεται στο άρθρο 12 ότι το Summit ε, συνέρχεται για να συζητήσει και όχι να αποφασίσει. Και νομίζω ότι είναι θετικό ότι στην τελευταία διευρυμένη ευρωομάδα σε μια συνάντηση έτσι κάπως χωρίς βεβαιότητα με ποιο καθεστώς συνεδριάζουν όπως τη Δευτέρα το βράδυ δεν είχαμε καμία αντίθετη άποψη για την αλλαγή αυτού του μέρους του άρθρου 12 και για το να υπάρξει μια πρόσκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς κανένα περιορισμό όχι, ότι θα έπρεπε να προσκληθεί. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει. Εντάξει, εμείς περιμένουμε κάτι τέτοιο. Θα ήταν κάτι το παράδεξο. Μετά από μια τόσο πλατιά συνένεση, το στοιχείο αυτό να μην αναφερόταν στο επόμενο προσχέδιο. Και το Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζει τη θέση των κρατών που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ. Το κάναμε και στο ψήφισμά μας και στην συνάντηση της Δευτέρας και θεωρούμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τόσο, ότι δεν είναι κατάλληλη η σημερινή διατύπωση μία, δύο φορές κάτι τέτοιο, τα όρους, όρια μάλλον, που δεν ταιριάζουν σε μια παρόμοια άτυπη συνάντηση και λόγω και της ερμηνείας που δίδεται σε αυτό το άρθρο. Βέβαια, αυτές οι βελτιώσεις από θεσμικής πλευράς που δεν ξεκαθαρίζουν το βασικό πρόβλημα μια συμφωνία κυβερνητική, αλλά τουλάχιστον ε, το ξεδοντιάζουν κάπως ε, στα πλαίσια αυτά. Εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, αμφιβολίες, επιφυλάξεις πολιτικές γιατί, γιατί ενώ εμείς προχωράμε με συγκεκριμένα γεγονότα για μια πειθαρχία ε, φορολογική. Προς το παρόν ακούμε μόνο λόγια για την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη, ενώ οι δύο πτυχές θα πρέπει να συμβαδίζουν και γι' αυτό το λόγο ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κατέθεσε τροπολογίες ε, για αυτό το θέμα στη συνθήκη και θα επιμείνουμε πέρα από τις συνθήκες ακριβώς στους κατάλληλους χώρους και με τις κατάλληλες διαδικασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνουμε τις επιλογές μας που αποτελούν προϋπόθεση για να πετύχουμε το στόχο που έθεσε όπως πρέπει ακριβώς και υπενθύμησε στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργό Δανία, ότι αυτή η πειθαρχία είναι απαραίτητη προπόθεση, αλλά όχι επαρκής για να προφυλάξουμε και το κοινωνικό ε, προφίλ και τις συμφωνίες, κάτι που άλλωστε θα εξασφαλίζαν και μια ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πάμε πέρα από τα φορολογικά θέματα, περιμένουμε τον ενεργό ρόλο που θα παίξει η Δανική Προεδρία ο πρόεδρος, ευχαριστώ Γκατιέρη και τώρα το λόγο βέβαια θα πρέπει να λάβουν όλοι οι συνάδελφοι. σα παρακαλώ λίγο συντομότεροι για να μπορέσει να απαντήσει όπως πρέπει και ο ε, Υπουργός ε, Χέφνερ, αλλά παρακαλώ σύντομα. herzlichen Dank. Uh, σας ευχαριστώ, θα μιλήσω αγγλικά για να πιο εύκολα. Θα ήθελα να εκφράσω μια μεγάλη ανησυχία, ένα μεγάλο φόβο που έχω, ότι προσπαθώντας να επιλύσουμε την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, θα φέρουμε την Ευρώπη σε μεγάλα προβλήματα. Αναπτύσσοντας στρατηγικές ε, διαδικασίες εκτός των συνθήκων, εκτός της κινητικής μεθόδου. Ολόκληρες γενιές πριν από εμάς ε, εργάζονταν για την κοινή Ευρώπη. Εργάζονταν για την ανάπτυξη των θεσμικών οργάνων, για την ανάπτυξη της δημοκρατικής βάσης που θα ενισχύσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα ερχόμαστε και αποδυναμώνουμε την κοινωτική μέθοδο, αποδυναμώνουμε το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή. Και δεν έχω πιστεί καθόλου ότι όλα αυτά είναι απαραίτητα και ότι θα επιλύσουν την κρίση. Άρα, αποτελούν τμήμα μίας λύσης, όχι όμως την κατεξοχήν λύση. Άρα σας ερωτώ. Τι θα γίνει μετά από το σημερινό δημοσιονομικό συμβόλαιο το οποίο συζητιέται για να επαναδομηθεί αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα της κοινή Ευρώπης με τρόπο ώστε να βασιστεί εκ νέου στη δημοκρατία, στην κοινωνική μέθοδο, στην διάκριση των εξουσιών, στη δυνατότητα των πολιτών να εκφράσουν την βούλησή τους μέσω των εκλογών, το οποίο συνεπάγεται να συμμετάσχει και το, και το κοινοβούλιο σε όλες τις διαδικασίες αυτές. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ερώτημα για όλους μας. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν στα πλαίσια της σημερινής ε, συνθήκης και τι πρέπει να γίνει πέρα από αυτήν για να καταλέξουμε σε ένα δημοκρατικό οικοδόμημα το οποίο θα ενσωματώσει την οικονομική και τη μισονομική συνεργασία η οποία είναι απαραίτητη ασφαλώς. Το επόμενο ερώτημα ή μάλλον πριν από το επόμενο ερώτημα θα ήθελα να τονίσω εκ νέου ότι θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα μας καθήκοντα αυτή τη στιγμή είναι να εμπλέξουμε εκ νέου και τους πολίτες. Γιατί αυτή τη στιγμή ο πολίτης κάθεται και παρακολουθεί αμέτωχος μία διαδοχή συνόδων και αποφάσεων στις οποίες ποτέ δεν συμμετείχαν και στις οποίες ποτέ δεν ακούστηκε η φωνή τους, ποτέ δεν ψήφισαν για το οτιδήποτε. Είναι απαραίτητο, αν δεν θέλουμε να χάσουμε αυτούς τους πολίτες από την Ευρώπη και αν δεν θέλουμε η Ευρώπη να διακατέχεται από ακροδεξιά αντιευρωπαϊκά κινήματα, να συμμετάσχει εκ νέου λοιπόν ο πολίτης. Και η εκκίνηση, η έναρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του πολίτη τον Απρίλιο, και το λέω ως ένας από τους συζητητές από πλευράς του Κοινοβουλίου, και ως ένα από τα άτομα που πρότειναν την ιδέα αυτή στα μέλη της συνθήκης της συνέλευσης πριν από δέκα έτη. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη λοιπόν η ευκαιρία για σας, για την Προεδρία από κοινού με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να καταδείξουμε στους πολίτες ότι είμαστε ανοιχτοί για τις ε, απαιτήσεις τους, για τις επιθυμίες τους για να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο εργαλείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα παρουσιαστεί αυτό το εργαλείο. Και είναι σημαντικό να το πάρουμε εμείς τα σοβαρά. Κάτι άλλο. Στο Ευρωπαϊκό Έτος του Πολίτη το 2013, το οποίο και προετοιμάζουμε σήμερα. Θα πρέπει να εξετάσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου περιλαμβάνονται, διαπιστώνω, πολλά καλά λόγια, αλλά συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες ενέργειες, το περιεχόμενο είναι ισχνό. Άρα θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία το έτος του πολίτη για να καταδείξουμε ότι η Ευρώπη ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή του πολίτη, του ενεργού πολίτη. Όχι μόνο για να διαφημίσουμε πόσο καλά τα κάνουμε όλα, αλλά για να ακούσουμε πραγματικά τις ανησυχίες, τις προτάσεις των πολιτών για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία. Προτιμάζω μια αγνομοδότηση από πλευράς της Επιτροπής μας για την πρωτοβουλία των πολιτών. Συναντηθήκαμε χθε με την Επιτροπή και μαζί με το Συμβούλιο θα πρέπει να εργαστούμε για μια καλύτερη διαμόρφωση του έτους του πολίτη. Και θα ήθελα να μου πείτε αν είσαστε ανοιχτό για μια τέτοια πρόταση. Τέλος, για το πρωτόκολλο της Αιχίας, να πω από πλευράς των Πρασίνων, με πάσα ειλικρίνεια, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, αυτό άλλωστε αποφάνθηκε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ισχύουν λοιπόν για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι θα ήταν παράδοξο και απαράδεκτο να δηλώνεται σε ένα πρωτόκολλο ότι αυτό δεν ισχύει απόλυτα για τον λαό της Τσεχίας, γνωρίζοντας ότι αυτό ποτέ δεν αποτέλεσε εκπεφρασμένη επιθυμία του τσεχικού λαού όταν ε, επικύρωσε το τσεχικό κοινοβούλιο, επικύρωσε και την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι άμεσα εκλεγμένοι του τσεχικού λαού ψήφισαν υπέρ της χάρτας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο κύριος Κλάους, ε, το γεγονός ότι βγήκε και υποστήριξε ότι δεν του άρεσε, ήταν περίεργο ήδη το ότι δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο. Αλλά δεν, είμαστε, δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος, δεν είμαι καθόλου μάλλον πεπισμένος ότι αυτό είναι προς το όφελος του λαού της Τσεχίας και της Ευρώπης. αμφισβητείται μάλιστα και στο ιστορικό της τσεχικής δημοκρατίας. Άρα θα προτείναμε να μην εξεταστεί το πρωτόκολλο. Ε, Ο συνάδελφος Νταφ το λόγο και μετά να δούμε και τους επόμενους ε, μια πρώτη απάντηση του Υπουργού και μετά ελπίζω να έχουμε το χρόνο να υποβάλλετε και άλλες ερωτήσεις. Μπρος Σόντεργκαντ. Ο κύριος Δάφ, θα είμαι όσο πιο λακωνικός γίνεται. Όπως είπατε, ε, δεν θα έχουμε την ε, χαρά να απολαύσουμε την παρέα σας και να συναντηθούμε σε μια συντακτική συνέλευση. Κάτι που φυσικά μας λυπεί ιδιαίτερος για τους γνωστούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει όμως θα ε, βρεθούμε για να συζητήσουμε τα θέματα των εκλογικών μεταρρυθμίσεων. Και ευελπιστώ ότι η έκθεση μου θα περάσει το Μάρτιο στην Ολομέλεια. Οπότε θα έχει την ευκαιρία η Δανική Προεδρία να εγκύψει το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο της Τσεχίας, όπως ξέρετε, είμαι εγώ εισηγητής για το θέμα αυτό και ακούσαμε τις απόψεις των συναδέλφων. Θα ήθελα να δηλώσω ότι η κατάσταση δεν είναι όπως παρουσιάστηκε στον ε, ψυχικό τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, ως μια επίθεση δηλαδή, του Κοινοβουλίου κατά του Πρόεδρου Κλάους. Εμείς απλώς προσπαθήσαμε να προασπίσουμε την κεραιότητα και να προωθήσουμε τη, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ισχύ του. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ανέκυψε το θέμα από τον κύριο Γκερέρο την, το γεγονό τη προσχώρηση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ECHR που είναι η προϋπόθεση για να, να γίνει υποχρεωτικός ο χάρτης. Ε, ε, χρειαζόμαστε να συντρέχει αυτή η προϋπόθεση, μάλλον το αντάλλαγμα για να ε, προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ECHR. Και αυτό ήταν συγκεκριμένο αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και είναι περίεργο που οι Βρετανοί είναι αυτοί που ακριβώς ανα, αναβάλουν τα πράγματα και περιπλέκουν την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Και μάλιστα διαβάζω στο Twitter ότι ο Πρωθυπουργό Κάμερον αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκφωνεί βαρισίμαντη ομιλία στο Στρασβούργο στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προσήλωση της Μεγάλης Βρετανίας στις αρχές των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ωραία όλα αυτά, αλλά ελπίζουμε ότι ε, αυτά τα λόγια να μετατραπούν και σε έργα, προκειμένου να εξασφαλιστεί συμφωνία και από τις 27 χώρες μέλη και το Συμβούλιο της Ευρώπης για την προσχώρηση στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώ... Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπω Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, υπάρχει μία πρόταση κάποια από τα συμβαλόμενα μέρη να προσπαθήσουν να συμπεριλάβουν μία δήλωση στη Νέα Συνθήκη προκειμένου να εκφράσουν την ελπίδα τους για πιο φιλόδοξα μέτρα προς την κατεύθυνση της ε, Δημοσιονομικής Φορολογικής Ένωσης. και δίνοντας ένα περιεχόμενο ε, στη συνθήκη αυτή, στο πακέτο αυτό, στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η προσέγγιση της Δανικής Προεδρίας ως προς την πρόταση αυτή που φαίνεται να κυκλοφόρησε, να αιωρείται τέλος πάντων στην ατμόσφαιρα στην Ιταλία και σε ορισμένες χώρες άλλες μέλη. Πιστεύετε ότι η νέα αυτή συνθήκη ε, θα περάσει πιο δύσκολα και θα καταστήσει ακόμη πιο διστακτική τη Δανία ως προς την προσχώρηση της στην Ευρωζώνη ή αντίθετα θα επισπεύσει αυτή τη διαδικασία. Ε, το λόγο έχετε εσείς κύριε Υπουργέ. Ξέρω λόγω πείρας ότι ο δύο συνάδελφοι σίγουρα επειδή είναι ιδιαίτερα περιληπτικοί θα είναι σύντομοι να τους αφήσουμε να λάβουν το λόγο και μετά να απαντήσετε. Μπρος. Παρακαλώ γρήγορα γρήγορα έτσι όπως περιμένω από σας άλλωστε. Okay. Right, you said... Uh, Είπατε, νομίζω ότι καλά άκουσα, ότι θέλουμε να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό έργο. Αυτά θα μπορούσε να τα είχε πει και η προηγούμενη προεδρία και η προπροηγούμενη δηλαδή. Και θα τα χρησιμοποιήσει και η επόμενη προεδρία κατά πάσα πιθανότητα. Δεν είναι ιδανική ατζέντα είναι η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έχει περάσει με μια διαφορετική α, σημαία. Είπατε ότι μια και είμαστε Προεδρία μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας θα έχουμε νομοθετικό ρόλο. Αλλά αυτό είναι ο λόγος του μιλητή και όχι του πολιτικού ηγέτη απαραίτητα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο de facto υπάρχει εδώ και δεκαετίες, αν και ουσιαστικά δημιουργήθηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας, πλέον έχει μόνιμο πρόεδρο που δεν είναι εκπρόσωπος κρατός μέλους και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του, του Συμβουλίου αυτού προεδρεύει η υπατή εκπρόσωπος η οποία ε, έλαβε αυτή την εντολή από ένα σώμα του οποίου ηγείται. Και έτσι τα κρατημέλη έχουν σημαντικά μικρότερες αρμοδιότητες. Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ότι πλέον είναι οργανωλικοί οι όροι. Όπως ε, διακυβερνητισμός, δεν ξέρω καν αν υπάρχει στο λεξικό αυτό, για να αναφερόμαστε σε αποφάσεις των κρατών μελών και αντίστοιχα κοινοτική μέθοδος για να αναφερόμαστε σε αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς τα κράτη-μέλη. Και αυτοί οι όροι χρησιμοποιήθηκαν σήμερα το απόγευμα. Μου προκάλεσε ενδιαφέρον από τα μέλη της Επιτροπής που άκουσα ότι θα καλέσουμε τους πολίτες να συμμετάσχουν πιο πολύ. Αυτό μου προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση και σε ό,τι αφορά τα σχετικά δημοψηφίσματα για τις συνθήκες. Λέτε δηλαδή ότι θα γίνουν σεβαστά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος αυτού και δεν θα διοργανωθούν δεύτερα δημοψηφίσματα. Γιατί φυσικά όταν μιλάμε για δικαιώματα του πολίτη, μιλάμε για το δικαίωμα του πολίτη να υπακούει σε εντολές. ευχαριστώ. Ο ε, τελευταία παρέμβαση. Θα ήθελα να μιλήσω στη γλώσσα μου για να μην <laughs> ταυτόχρονα να μην πείτε ότι δεν υπάρχει συνεννόηση με τον Υπουργό. Θα πρέπει να δούμε αν χρειάζεται κοινοτική μέθοδος ή διακυβερνητική, να δούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε στις συμφωνίες ε, ευρωπαϊκής ε, Και όπως είπε και ο Υπουργό ε, στην παρέμβασή του, θα πρέπει να αναφερθούμε στο άρθρο 48 η παραδοσιακή διαδικασία αναθεώρησης, μήπως θα πρέπει κανείς να προσφύγει στην ε, διαδικασία απλοποιημένης επικύρωσης. Ε, τι παρατήρησα ότι ο Υποργό, ε, ακριβώς επειδή δεχτήκαμε εμείς τις δύο πρώτες περιπτώσεις την απλοποιημένη διαδικασία μας ευχαρίστησε. Εδώ πρόκειται για μικρού βεληνικούς θέματα ε, εντάξει, η πρώτη περίπτωση ήταν το θέμα της διεύρυνσης, ε, της σύνθεσης του Κοινοβουλίου και με πολλά νέα μέλη και την δεύτερη αναθεώρηση ήταν κάπως σημαντικότερη βέβαια, αλλά τέλος πάντων ε, χρειαζόταν να εξετάσουμε τα πράγματα στα γρήγορα και θα ήταν ε, διαφορετικά τα πράγματα αν είχαμε την παραδοσιακή διαδικασία. Ξέρω πως τίθεται το πρόβλημα, τι γίνεται. Πότε εμεί όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συνήθη διαδικασία, την παραδοσιακή που προβλέπουν ε, πολλέ συνθήκε. Όχι είναι για μικρά πράγματα γιατί να πείτε κάτι τέτοιο και όχι γιατί όταν είναι σημαντικά, αλλά επειδή Ευρωπαϊ... για θέματα ευρωπαϊκή οικονομία, επειδή δεν έχουμε χρόνο να καθυστερήσουμε. Τι γίνεται λοιπόν. Ε, Αυτή είδαμε το πρόβλημα στο Ευρωμαρόμετρο που δείχνει ακριβώ ότι ε, είναι ομοιεμένη η δημοτικότητα ακριβώ η δικιά μας από τη στιγμή που δεν επιφέρουμε λύσεις για να ξεφύγουμε από τα προβλήματα αυτά, να τα λύσουμε. Είχαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας για να, για να πούμε για μια δημοκρατική διαδικασία στα πλαίσια της μεταρρύθμισης των συνδικών. Και ακόμα κάτι ακόμα. Μας είπε ο Υπουργός ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στη συμφωνία αυτή περί και αυτή είναι θέση της κυβέρνησης και με την υποστήριξη δηλαδή ακριβώς του Κοινοβουλίου του, της Δανίας αλλά εκεί μπαίνουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Μπορεί να μας επιβεβαιώσει Μάλλον όχι. Ο υπουργό ότι συμπεριλαμβάνεται κάτι στο Δανικό Σύνταγμα που να εμποδίζει τη Δανία να υπογράψει οποιαδήποτε έκδοση του Συμφώνου για τον προϋπολογισμό και πού να είναι στην τράπεζα, εντάξει, καμία εκδοχή. Εδώ το πράγμα που απαιτείται ποιο είναι, ένα δημοψήφισμα. Και αναρωτιέμαι, θεωρεί ο υπουργό ότι μπορεί να συμμετάσχει η Δανία, αλλά αποφεύγοντα ένα δημοψήφισμα, γιατί νομίζω ότι θα ήταν ε, αρνητική ένδειξη και απέναντι στην ελληνική για του συναδέλφου, γιατί μιλάμε για την ελληνική. Εάν θεωρούμε ότι είναι κάτι το σημαντικό αυτή η ελληνική, τότε θα προχωρήσουμε πραγματικά σε βάθο και να θέσουμε ίσω το θέμα ακριβώ στου εκλογεί, αν θεωρούμε ότι κάτι το σημαντικό. Αλλά το ερώτημα ποιο είναι, τι γίνεται. Είναι σημαντικό από τη στιγμή που αποφεύγουμε μια δημοψήφισμα. Έτσι είναι τα πράγματα. Ευχαριστώ, λέω ο πρόεδρο. Ε, ολοκληρώσαμε με τι ε, πολλέ και διάφορε παρεμβάσει. Ε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις απορίες σας και να θίξω όλα τα ζητήματα που επισημάνατε κι εσείς. Ο κ. Σταρκόφσκι είπε ότι χαίρεται για τη θετική νότα και γενικώ ε, την θετική διάθεση της Δανικής Προεδρίας. Θα ήθελα να σας πω ότι διανύουμε την ε, βαθύτερη κρίση στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Κάτι που μας ε, φορτώνει τεράστια ευθύνη. Κοινή ευθύνη όμως του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει από κοινού να την επομισθούμε. Και σίγουρα αυτή δεν είναι καιρή για θεσμικούς ε, διαπληκτισμούς και θεσμικές αντιπαραθέσεις. Είναι δύσκολη καιρή, γι' αυτό καλό είναι να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Και βλέπετε τη Δανική Προεδρία σαν γέφυρα σε ταραχμένα νερά, αλλά είδατε ότι με το δημοσιονομικό πακέτο ακόμη δεν μπήκαμε, δεν αρχίσαμε να περπατάμε πάνω στη γέφυρα. Και είπατε ότι ίσως είναι πρόωρο να προεξοφλούμε την έκβαση διαπραγματεύσεων που δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να προτρέχουμε. Αλλά είπα ότι από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα δημιουργείται μια αισιοδοξία ότι θα βρεθεί μια τελική λύση που θα είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά και εσείς αλλά και οι συναδελφοί σας ρώτησαν ποια είναι η ιδανική θέση στο θέμα αυτό. Εμείς έχουμε ένα opt-out, ρήτρα αυτοεξαίρεσης για το, για το ευρώ. Και σίγουρα θα το λάβουμε υπόψη. Δεν πρόκειται να συμμετέχουμε αν υπάρχει μια αντίφαση ε, με, το, με τη ρήτρα αυτοεξαίρεση. Αυτή είναι η θέση της πλειοψηφίας ε, της κυβέρνησης και της Δανικής Βουλής. Τώρα, το θέμα του συνταγματικού ισοδύναμου νόμου. Πρόκειται για μια συζήτηση που συνεχίζεται μεταξύ Δανίας και άλλων χωρών. Γιατί στη Δανία ισχύει ένα ιδιάζον σύστημα που δυσκολεύει κάπως τα πράγματα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Αλλά είναι μία από τις εκκρεμότητες που σας επισήμανα προηγουμένως. Πάντως, αυτός δεν είναι ο πρωταρχικός ρόλος της Προεδρίας. Θα είναι μια συμφωνία, μια συνθήκη μεταξύ των χωρών μελών. Και σε αυτό το πλαίσιο γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Και όπως είπατε και εσείς, πρόκειται για μια ιδιάζουσα κατάσταση στο κοινοτικό σύστημα, στο ευρωπαϊκό σύστημα, γιατί δεν είναι ο συνήθις τρόπος διαθέτησης των πραγμάτων και ανέβρεση συμφωνιών. Είναι μια πρόκληση, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε λύση. Και ως χώρα μέλος, αλλά και ως Προεδρία φροντίσουμε να βρεθεί λύση και ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Ο Ερίκε έθεσε μερικές ερωτήσεις και κάνει και πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Ένα θέμα που τέθηκε από πολλούς αφορούσε το πρωτόκολλο της Ιρλανδίας και της Τσεχίας. Καταλαβαίνω για... γιατί γίνεται συζήτηση. Καταλαβαίνω τις απόψεις ό,τι αφορά τη συζήτηση για την Τσεχία. Αλλά θα πρέπει να σημειώσω και το εξή. Εκτός κι αν η τσεχική κυβέρνηση ζητήσει από όλου μα. το ζητήσει από όλου μα, θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να ανταποκριθούμε στις υποσχέσεις του 2009 που διασφαλίζουν ότι, που διασφάλισαν ότι τέθηκε σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας. Είτε συμφωνούμε είτε όχι με τα θέματα της τσεχικής ε, δημοκρατίας. Αυτό ήταν που υποσχεθήκαμε στην τσεχική δημοκρατία και άρα μας δεσμεύει αυτή η υπόσχεση με ότου ε, επιθυμήσει το αντίθετο ο λαός της Τσεχίας. Και αυτό θα είναι ο τρόπος που θα συνεχίσουμε το έργο μας. Επίσης, τέθηκε το θέμα των ανθρωπινών δικαιωμάτων, το οποίο έθιξε και ο κύριος Νταφ αλλά και άλλοι. Η ιδανική κυβέρνηση τονίζει ιδιαίτερα την προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων και θεωρεί πολύ θετικό βήμα την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χάρτα των ανθρωπινών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και η Δανία θα εργαστεί σκληρά για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων θα αποτελέσει αυτό υψηλή προτεραιότητα της Δανικής Προεδρίας. Δεν αναμένουμε ωστόσο οριστική διαπραγμάτευση στον τομέα αυτό, αλλά θα αποτελέσει προτεραιότητά μας. Θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε το, το γρηγορότερο δυνατόν. Επίσης, τα ερωτήματα για την έκθεση Μάρτιν. Όπως είπα, είναι πρώιμη η φάση. Αλλά δεσμευόμαστε για να βρούμε λύσεις. Θα ήθελα να απαντήσω και στα λόγια του Προέδρου και άλλων, αν είναι δυνατή η εξέβρεση λύση, τότε ο Φεβρουάριος δεν αποτελεί ουτοπικό σενάριο. Θα ήταν ωφέλιμο για την Προεδρία να γίνει η ψηφοφορία σε μετέπειτα χρονική στιγμή, μετά το Φεβρουάριο. Παράλληλα, να σας πω ότι σκοπός και πρόθεση της πρότασής μου δεν είναι να καθυστερήσω την απάντηση, αλλά να δώσουμε χρόνο για να βρεθεί κοινό τόπος για συμβιβασμό. Και φυσικά θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Μάρτιν όταν θα ξαναέλθει στο Κοινοβούλιο. Αλλά θα ήθελα επευκαιρίας να σας ε, ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας και για τις προσπάθειές σας στο πλαίσιο αυτό. Τέθηκε στη συνέχεια το ερώτημα των ε, εξουσιών των διερευνητικών. οι αρμοδιότητες ε, των κοινοβουλίων διαφέρουν σημαντικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, άρα δεν υπάρχει σημείο σύγκριση. Επίσης, η Ένωση, παρά το γεγονό ότι έχει πολλές αρμοδιότητες σε πολλούς τομείς, δεν συγκρίνεται με ένα κράτος μέλος σε ό,τι αφορά την αρχή της εκχώρησης και έτσι δεν μπορεί να ξεπεράσει τις αρμοδιότητες που τις εκχωρούνται από τις συνθήκες. Αυτό ασφαλώς αποτελεί ένα από τα θέματα που προκαλούν πολλές συζητήσεις και έχουμε σημαντικό δρόμο να διανύσουμε μπροστά μας, αλλά προσβλέπω σε αυτές τις συζητήσεις. Ύστερα, ο κύριος Γκουατιέρη έκανε κάποιες πολύ σημαντικές παρατηρήσεις για το ρόλο του Κοινοβουλίου και το πώς θα συνεργαστούμε. Θα είμαι ειλικρινή μαζί σα. Εμεί θα θέλαμε από πλευράς Ιδανική Προεδρία μία συμφωνία στην οποία θα συμμετείχαν και τα 27 κράτη-μέλη. Αυτό θα αποτελούσε το καλύτερο, την καλύτερη λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινωτική Μέθοδο, που θα έδινε ένα καθημερινό χαρακτήρα στα πάντα. Αυτό δεν ήταν δυνατόν. Άρα θα πρέπει να βρούμε πλέον μία λύση υπό δύσκολους όρους. Είναι ελπίδα και επιθυμία μου και της Δανικής Προεδρίας να εξεύρουμε λύσεις. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τερματίσει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία αυτή για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Κατανοώ ιδιαίτερα τις απόψεις που εκφράστηκαν ως προς αυτό και επίση καταναμώ και την επιθυμία των κρατών μελών εκτό Ευρωζώνη που θα θέλανε να συμμετάσχουν στι συναντήσεις για την οριστική διαμόρφωση του Δημοσιονομικού Συμβολέου. Ο κύριος Χέφνερ ανέφερε ότι θα ήθελε η Δημοσιονομική Σύμβαση να αποτελέσει το συντομότερο δυνατόν τμήμα του κανονικού ευρωπαϊκού συστήματος. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ λογική και σωστή προσέγγιση και αυτό αναμένω ότι θα συμβεί. Τώρα με ποια ταχύτητα και σε ποια χρονική ε, στιγμή αυτό θα το δούμε. Αλλά αυτό είναι ο απότερος στόχος. Επίσης σημαντικό είναι, συμφωνώ, να μην αρχίσουμε να δημιουργούμε θεσμούς και θεσμικά όργανα, αλλά να βρούμε μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα μας επιτρέπει να λαμβάνουμε τις απαραίτητες αποφάσεις χωρίς ε, να χρειάζεται να λαμβάνονται νέες πρωτοβουλίες. Μετατέθηκε το θέμα της συμμετοχής των πολιτών. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και εσάς και όσους ε, συνεργάστηκαν για να πετύχουν πρώτο στον τομέα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, η πρωτοβουλία των πολιτών να αποτελέσει ένα τρόπο με τον οποίο ο κοινό θνητός, ο καθένας από τα 500 εκατομμύρια, να μπορεί να θέσει την ατζέντα του, χωρίς να είναι επίτροπος, χωρίς να είναι υπουργός, χωρίς να είναι ευρωβουλευτής να μπορεί όμως να επηρεάσει αυτά που συμβαίνουν εδώ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό και σίγουρα θα ήθελα να συναντηθούμε και να συζητήσουμε την ε, ατζέντα του επόμενου έτους και ελπίζω να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. Ο κύριος Νταφ ε, μίλησε για τα θέματα αυτά. Είναι πάντα χαρά μου όταν τα προσεγγίζουμε και ήδη υπέβαλε κάποιες παρατηρήσεις. Σε ό,τι φορά την έκθεσή του, την έκθεση DAF, φυσικά σέβομαι το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και περιμένω με αδημονία τη συζήτηση που θα λάβει η χώρα. και όταν ξέρουμε και την έκβαση της ψηφοφορίας, ξέρουμε και τι μας περιμένει. Σας το είπα και στην Κοπενχάγη. Δεν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ε, άμεσο θέμα η αναθεώρηση της συνθήκης. Πάντως καταλαβαίνω για ποιο λόγο αναλάβατε τη σχετική πρωτοβουλία και ξέρω ότι πάντα οι εκθέσεις σας είναι, χαρακτηρίζονται από μεγάλο επαγγελματισμό, από την προσήλωση στα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και οι δύο γνωρίζουμε θαυμάσια ότι το θέμα δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα έχουμε πάντως την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ανέφερα και προηγουμένως και ευελπιστώ ότι θα βρούμε λύση και εκεί. Κύριε Μπρόγκ, είπατε ότι άλλαξα τα πράγματα με τις ε, εκπεριτροπής προεδρίες. Οι προεδρίες δεν είναι αυτό που ήταν. Όντως, υπάρχουν αλλαγές. Πάντως η Ιταλική Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανταπεξέλθει στις ε, ευθύνες, να μην διαψεύσει τις προσδοκίες και να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ύψης προτεραιότητες της δικής μας Προεδρίας. Αυτό το αναφέρατε πολλοί από εσά και φυσικά είναι και σημαντική προτεραιότητα δική μας. Και προσβλέπουμε σε υποστήριξη δική σας αυτή την προσπάθεια. Ο κύριος Σόντεργκορτ μου έθεσε την ερώτηση στα Δανέζικα και εγώ θα απαντήσω επίσης στα Δανικά. Για να με κατανοήσει και εκείνος όπως ε, εκείνος ζήτησε να έχουμε απευθείας επικοινωνία. Γι' αυτό παρακαλώ να δεχτείτε αυτή την σύντομη δανεική ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Σαντεργόρτ, είπατε ότι ε, υπάρχει πλειοψηφία στη Δανική Βουλή που είναι υπέρ αυτού του δημοσιονομικού συμφώνου. Και είπε ότι σέβεται αυτή την πλειοψηφία και έθεσε μία ερώτηση για την οργάνωση και διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος. Ως προς αυτό η δανεική κυβέρνηση είναι σαφής. Το άρθρο 20 του Δενικού Συντάγματος μιλάει ότι σε, λέει ότι σε περίπτωση ε, που τίθεται ζήτημα κυριαρχίας θα πρέπει ε, να διοργανωθεί δημοψήφισμα εκτός αν υπάρχει αντίθετη γνώμη του, των πέντε εβδόμων της ε, Δανικής Βουλής. Η θέση του κόμματος του κυρίου Σέντεργκαρτ είναι κατά αυτής της θέσης, αλλά ε, δεν συγκεντρώνει την πλουσία των πέντε εβδόμων. Από τη στιγμή που δεν πρόκειται για θέμα κυριαρχίας, οπότε είναι υποχρεωτικό το δημοψήφισμα, εναπόκειται στη Δανική κυβέρνηση να λάβει απόφαση για την ε, ε, συμμετοχή της Δανίας. Άλλωστε η πλειοψηφία της ε, Δανικής Βουλής είναι υπέρ αυτής της θέσης και χαίρομαι ως υπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων για την σημαντική αυτή υποστήριξη της Δανικής Βουλής. Πάντως άσχετα με το αποτέλεσμα μπορούμε να συνεχίσουμε με τον Σέρεν Σάντεργκαρτ για τα υπέρ και τα κατά της πιθανής δανικής συμμετοχής στο μέλλον. Πάντως, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί είχα την ευκαιρία ε, να λάβω μέρος σε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Συνεχίζω λοιπόν στα δανεικά μια και ξεκίνησε. Νομίζω ότι σημαντικό είναι να συζητάμε άσχετα με το σε ποια γλώσσα γίνεται η συζήτηση. Ναι, ήδη την Κυριακή που μας έρχεται και εγώ θα είμαι παρόν, αλλά και άλλο μέλη της Επιτροπής ε, θα είμαστε στην Κοπενχάγη. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να συνεχιστεί ο διάλογος. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και θα συνεχίσουμε για λίγη ώρα ακόμα τις εργασίες μας στην Επιτροπή μας. Allora. Για να δούμε, για να δούμε. Ξανά στις εργασίες μας που είχαμε διακόψει στην εκλογική διαδικασία. Ο κύριος Νταφ. Εντάξει, με ακούτε. Λοιπόν, ε, εκλογική διαδικασία. Είχαμε ακόμα την κυρία Γιαννάκου και Ταρκόφσκι. Η κυρία Γιαννάκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Νταφ για τη δουλειά που έχει κάνει παρά το γεγονός ότι η έκθεση του προκαλεί σοβαρές διχογνωμίες. Ε, κύριε Πρόεδρε, ιδιαίτερα στο σημείο που αφορά στην ανακατανομή των εδρών, βεβαίως γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί απόφαση του Συμβουλίου. Αλλά νομίζω ότι είναι η πλέον ακατάλληλη στιγμή να εμφανιστεί το Κοινοβούλιο ζητώντας μια ανακατανομή των εδρών υπέρ των μεγάλων χωρών. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η προσήλωση στο κοινοτικό δεδομένο, στον κοινοτικό τρόπο λειτουργίας και σκέψης, οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν υπάρχει απόλυτη αναλογικότητα στην εκπροσώπηση ούτε στο Κοινοβούλιο, ούτε στο Κορεπέρ με τις ψήφους και αυτό ακριβώς εξασφαλίζει το να μην μπορούν οι μικρές χώρες να απειλήσουν τις μεγάλες ούτε και αντιστρόφως. Ε, κάθε αλλαγή υπέρ των μεγάλων χωρών ή υπέρ της αναλογικότητας κύριε Πρόεδρε σημαίνει επιστροφή στο διακυβερνητισμό. Τότε με αυτή τη λογική δεν υπάρχει κανένας λόγος για τις μικρές ή μεσαίες χώρες να δεχτούν διαδικασίες με αποφάσεις πλειοψηφίας. Έχω την εντύπωση και θέλω να το πω στον κύριο Νταφ ότι είναι η χειρότερη εποχή για μια τέτοια προσέγγιση. Θα δημιουργήσει ε, αυτό δημοσιευόμενο και εμφανιζόμενο στα μίντια θα δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις στις μεσαίες χώρες από τις οποίες στην ουσία ζητείτε να αφαιρεθούν έδρες και θα ενισχύσει τον ευρωσκεπτικισμό. Επίσης κύριε Πρόεδρε, η υπόθεση της κατανομής δυνάμεως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολιτική υπόθεση. Δεν είναι υπόθεση μαθηματικού τύπου. Σε καμία περίπτωση. Τα μαθηματικά είναι μια ανελαστική επιστήμη. Εγώ ως επαγγελματίας είμαι των θετικών επιστημών που σου δίνει απαντήσεις ανάλογα με αυτά που ρωτάς. Εάν κάνεις λάθος ερωτήσεις βεβαίως δίνονται λάθος απαντήσεις. Δεν είναι δυνατόν να υπολογίζονται οι έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μαθηματικό τύπο. Και δεν είναι δυνατόν συνάδελφοι που ανήκουν σε κράτη-μέλη που υποτίθεται ότι θα πάρουν περισσότερες έδρες να θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι απλό και μπορεί να αποφασιστεί έτσι επειδή θα εξασφαλιστεί μια πλειοψηφία θέλω κύριε Πρόεδρε να σας πω ότι το θέμα του πότε θα οριστούν οι ευρωεκλογέ βεβαίως είναι θέμα μιας οποιασδήποτε απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η λίστα η πανευρωπαϊκή δεν βρίσκει σύμφωνες ορισμένε πολιτικές ομάδες αλλά ιδιαίτερα για αυτό που αφορά στο μαθηματικό τύπο θέλω να σας πω ότι κάθε προσπάθεια να λειτουργήσει το βάρος των αποφάσεων υπέρ των μεγάλων χωρών θα αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της Ευρώπης που εμείς πιστεύουμε. Θα δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις στις μεσαίες χώρες ε, και βεβαίως ε, το Συμβούλιο θα αποφασίσει αλλά δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να εμφανίζεται το Κοινοβούλιο με τέτοιες απόψεις. Τότε ε, ποια επίκληση κύριε Πρόεδρε κάνουμε περί ολοκλήρωσης της Ευρώπης, περί εφαρμογής συνθήκης της Λισαβόνας λοιπά... Όταν απλώς ο καθένας ζητάει να πάρει όλο και περισσότερα. Και αυτό είναι εις βάρος επαναλαμβάνω της κοινοτικής λογικής. Αλλιώς να λειτουργήσουμε όλοι σε διακυβερνητική λογική και να παίρνονται αποφάσεις με ομοφωνία. Για να γνωρίζουμε όλοι μας ότι έχουμε εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο και τα θέματα της εθνικής μας κυριαρχίας. Εγώ δηλώνω κύριε Πρόεδρε ότι θα καταψηφίσω, λυπάμαι που θα το κάνω, θα καταψηφίσω την έκθεση του κυρίου Νταφ στο βαθμό που μένει με αυτή την άποψη ή στο βαθμό που οποιαδήποτε τροπολογία έχει υποβληθεί από οποιονδήποτε, από οποιαδήποτε πολιτική ομάδα εγώ προσωπικά θεωρώ ότι υπονομεύει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιαννάκου, σας ευχαριστούμε γιατί σαφώς ε, αναλύσατε ποια είναι αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται εδώ όταν μιλάμε για τον εκλογικό νόμο. Ο κύριος Σταρκόφσκι. I didn't ask for the floor. Our position was Δεν ζήτησα το λόγο. Την θέση μας την παρουσία ο σκιώτης μας και δεν πρόκειται να επαναλάβω τις απόψεις του. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο και όσοι έμειναν για να ακούσουν και την απάντησή μου. Νομίζω ότι ο Τζέραλτ απάντησε με επιτυχία στο θέμα το οποίο έθεσε ο κύριος Σουέπφλινγκ για την πίεση στις μεσαίου μεγέθους χώρες και ως προς τον αντίκτυπο που θα έχει σε αυτές ενός μαθηματικού τύπου, ένας μαθηματικός τύπος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι, διαφόρων ειδών τύποι και είμαι βέβαιος ότι θα είναι δυνατόν μετά από έρευνα του θέματος αυτού και με μαθηματικούς κατά την ε, έναρξη της Επιτροπής να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία λίγο πολύ θα είναι ικανοποιητική για όλους. Και αυτό ανταποκρίνεται στα κριτήρια της συνθήκης σε ό,τι αφορά το κριτήριο της, ε, της, φθήνουσας, της αναλογικότητας. Και θα ανταποκρίνεται και στα, στις καταγγελίες που λάβαμε από το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Θα ήθελα να ζητήσω από αυτούς που αρνούνται να εξετάσουν τη, βιωσιμότητα ενός μαθηματικού τύπου, τι ε, έχουν να προτείνουν. Η κυρία Γιαννάκου δεν μας είπε τι έχει να προτείνει, ποια είναι η δική της πρόταση για να συμπεριληφθούν κάποια μέλη από την Κροατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά το 2014 λέει ότι το status quo θα πρέπει να παραμείνει πάντα για ίδιο, το ίδιο για την Ελλάδα ή μήπω λέει ότι το μέγεθος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να αυξηθεί και μάλιστα εκθετικά προκειμένου τα καινούργια κράτη και είναι πολλά τα καινούργια κράτη στα Δυτικά Βαλκάνια ενδεχομένως, που θα προσχωρήσουν. Προκειμένου λοιπόν και αυτά τα νέα κράτη-μέλη να έχουν και αυτά ευρωβουλευτές να ξεπεράσουμε τους 751. Και αυτό θα ήταν κατά παράβαση της συνθήκης. Δεν κατανοώ. Κατανοώ μάλλον τους φόβους που εκφράζονται για την απώλεια εδρών, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να μην υπάρχει μια επικοδομητική ε, διάθεση για την εξαπλήση λύσης. και νομίζω ότι η πλειοψηφία του ΕΛΚ θα ακολουθήσει την σοφή σύσταση των σκιωδών και θα αποτελέσει επικοδομητικό μέλος των συζητήσεων. Ο κύριο Γκουαλτιέρη είπε ότι δεν του αρέσει το ότι υποστηρίζω τον κατάλογο ψηφοφορίας στην ε, τροπολογία 31 και ότι γι' αυτό μπορεί να αντιταχθεί σε αυτήν. Νομίζω ότι συμφωνεί ωστόσο μαζί μου ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την τροπολογία του κυρίου Βίλαν, την 30, για την ημερομηνία. για το χρονοδιάγραμμα λήψης αποφάσεων σε ό,τι αφορά την ημέρα των εκλογών. Νομίζω ότι προτείνει να αρχίσει η παράγραφος 4 με τη λέξη αποφασίζει και θεωρεί ότι αυτό καθορίζει. Θεωρεί ότι η διατύπωση αυτή δεν είναι αρκετά επιτακτική, αλλά το determines είναι πολύ πιο αυστηρό από ότι το proposes, προτείνει. Άρα, δεν θα ήθελα να αποδυναμωθεί η διατύπωση. Δεν θα ήθελα να μπει η λέξη proposes, προτείνει. Αν θεωρούμε ότι θα πρέπει να αλλάξει η διατύπωση. Και αυτό υποστηριχθεί από την πλειοψηφία. Φυσικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για τους λόγους που ανέφερε ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα σημεία επί της ουσίας. Και προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία. Θα πρέπει να αρχίσουμε με τη συνάντηση των συντονιστών. Κάτι όμως σύντομα, σύντομα η κυρία Γιαννάκου. Κύριε Πρόεδρε, καμία σχέση δεν έχει η πρόταση του κυρίου Νταφ με την είσοδο της Κροατίας ή άλλων κρατών μελών. Η έκθεση του κυρίου Νταφ προτείνει ένα μαθηματικό τύπο ο οποίος θέλει να ενισχύσει ορισμένες μεγάλες χώρες. Εγώ δεν προτείνω να αυξήσουμε τον αριθμό των μελών, να μείνουμε στο 751 που ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνας. Κάθε φορά που μπαίνουν νέες χώρες θα γίνει ανακατανομή σε συνεννόηση με το Συμβούλιο. Παραδείγματο χάρη η χώρα μου είχε 25 βουλευτές και σήμερα έχει 22. Αλλά ο μαθηματικός τύπος του κυρίου Νταφ θέλει να αφαιρέσει τεράστιο αριθμό βουλευτών από τις μεσαίες χώρες και να τις δώσει σε συγκεκριμένες χώρες. Λοιπόν, κύριε Νταφ, ξέρετε πόσο σας σέβομαι και σας εκτιμώ, αλλά καμία σχέση δεν έχει η έκθεσή σας με την, αύξηση, με την ανακατανομή που πρέπει να γίνει <clears throat> για την είσοδο της Κροατίας ή άλλων κρατών μελών. Αυτό είναι μια τελείω άλλη υπόθεση που θα αποφασιστεί κάθε φορά τόπου, πάλι με κριτήριο την κοινοτική λογική ή την κοινοτική πολιτική. Ευχαριστώ. Yes. Yeah. Yeah. I, I would only ask uh, Mrs. Απλώς να ρωτήσω την κυρία Γιγανάκου, την οποία σέβομαι πλήρως. Θα ήθελα να την παρακαλέσω μάλλον να διαβάσει πολύ προσεκτικά τη συμβαστική τροπολογία Γ. Εκεί αναφέρω ότι πρέπει να εγκαινιάσουμε διάλογο με το Συμβούλιο και φαντάζομαι συμφωνεί μαζί μου. Διάλογο λοιπόν με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την ε, αναθεώρηση της πράξης αυτής και μιλώ για την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας σε ό,τι αφορά την ανακατανομή των εδρών στα πλαίσια της αρχής της φθήνουσας αναλογικότητας. Δεν προτείνω ένα συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο. Δεν προτείνω κανένα τύπο εγώ. Απλώς λέω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε συζήτηση για ένα τύπο στις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο. Μπορεί σε τελική ανάλυση να έχει δίκιο κύριε Γιαννάκου και να ασφάλω εγώ. Ότι να μην είναι δυνατό δηλαδή να καταλήξουμε στη συμφωνία για ένα τύπο. Οπότε θα πρέπει να επανέλθουμε στην παλιά διαδικασία. Ε, αλλά αυτή η διαδικασία του να δώσουμε μάχη για τις έδρες δεν είναι και πολύ νομότυπη. Εντάξει, κλείνει εδώ η συνάντηση της Επιτροπής μας. Ε, μια στιγμή να διακόψουμε και αμέσως αρχίζουμε και πάλι με τη συνάντηση των συντονιστών. Τρία λεπτά διακοπή ώστε να μπορέσουν να αποχωρήσουν όσοι δεν είναι συντονιστές.